Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε και ξεκινάμε με μία δημόσια ακρόαση η οποία αφορά στην ε, χρήση της τεχνητής νοημοσύνης ε, στον εκπαίδευση και τον πολιτισμό και τον οπτικοακουστικό τομέα. Έχουμε διάφορους ε, καλεσμένους, γι' αυτό θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, έτσι ώστε να έχουμε χρόνο για κάθε παρουσίαση η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόν εδώ τον τομέα σπάνια συζητιέται. Οι μεγάλες λεπτομέρειες δεν μας είναι γνωστές, έχει, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει μια σοβαρή πολιτική συζήτηση για αυτό το θέμα. Ε, είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς επηρεάζει τα σχέδια μαθήματος, ε, την παραγωγή ταινιών. Είναι ένα θέμα λοιπόν μεγάλης σημασίας ε, και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να μάθουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, ειδικά εφόσον ο τομέας αυτό, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει αυτόν τον τομέα και να υπάρχουν και ρυθμιστικές επιπτώσεις στον επόμενο το επόμενο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα έρχονται πιο γρήγορα από ό,τι κανείς περιμένει. Και ήδη σήμερα μιλάμε για θέματα όπως τα deep και άλλα ε, κρίσιμα ζητήματα Οπότε υπάρχει από τη μία πλευρά μια τεράστια ευκαιρία να συνδεθούμε με την τεχνητή νοημοσύνη, από την άλλη όμως ε, καλό είναι να ξέρει κανείς τι κάνει και τι επιπτώσεις αυτό θα έχει. Είναι πολύ σημαντικό για μας ε, να ρίξουμε φως στις διάφορες πτυχές αυτού του θέματος. Έτσι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη είναι μία από τις προτεραιότητε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την νομοθετική περίοδο και η δική μας Επιτροπή του επόμενου μήνε θα ασχοληθεί εντατικά με αυτό το θέμα. Θα υπάρχει μία ήδη έκθεση πρωτοβουλία για το θέμα των οπτικοακουστικών. Υπάρχουν γνωμοδοτήσει, αλλά και άλλε εκθέσει από τη Γιούρη και τη Λίμπε βρίσκονται σε επεξεργασία. Ε, σε αυτέ λοιπόν ε, εξετάζονται τα διάφορα στοιχεία της κάθε επιτροπής. Έχουμε τρία μέλη, μέρη στην ε, ε, ακρόαση αυτή. Θα μιλήσουμε για την εκπαίδευση, τις γλώσσες κτλ. Θέλουμε να έχουμε Επίσης, να, τις προοπτικές, να δούμε ακριβώς στον τομέα του πολιτισμού ποιες θα είναι οι επιπτώσεις συγκεκριμένα στα απτικοακουστικά, έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις ε, προκλήσεις και να δούμε τι θα γίνει όταν πλέον εφαρμοστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Θα υπάρχει μια παρουσίαση για το deepfake, θα έχουμε εικόνες τεχνητής νοημοσύνης ε, και ακουστικά στοιχεία τα οποία αλλάζουν την εικόνα. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα εξετάσουμε και να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Χρειαζόμαστε τις πληροφορίες ε, από τους ειδικού και εμπειρογνώμονες ε, που θα μοιραστούν μαζί μας τα όσα γνωρίζουν για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ξεκινάμε με τον Αντρές ε, Βασίλειευς, που είναι ο Διεθνός Σύμβουλος του TILDE και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Big Data Value Association και του BDVA Public Private Partnership Board. Επίσης έχουμε τον κυρία Ντόρα Ματαβοζόφσκη Φίλιπ, η οποία είναι project leader της ομάδας εργασίας για την εκπαίδευση στην ε, Συμμαχία της Τεχνητής Νοημοσύνης της Ουγγαρίας και τέλος έχουμε την κυρία Λεωνόρα Ροζάτη, ε, η οποία είναι ε, δικηγόρος, καθηγήτρια ε, στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, ο δόκτωρ Κρίστοφ Κρόνκε, που είναι postdoc fellow στον δημόσιο δίκαιο στο Ludwig Maximilian Universität του Μονάχου και τον Μάικλ Κόλτβεϊ από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα για την Τηλεόραση και τον Κινηματογράφο στο Μόναχο. Έχετε ο κύριος Αντρέης Βασιλεύσκη έχει πρώτος το λόγο για 10 λεπτά. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, θέλω να, αναφέρω, να αναφερθώ στο θέμα αυτό. τι προκλήσεις μπορεί να μας δημιουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη και σε σχέση με τον πολιτισμό και την παιδεία. Θα περιγράψω κροθυγός τις εξελίξεις εν γέννη, δεντολογικά θέματα, ηθικά θέματα, που απορρέουν από τεχνητή νοημοσύνη, ο ρόλος του πολιτισμού, της κουλτούρας σχετικά με αυτό και μετά προβλήματα που παρουσιάζονται όσον αφορά τη γλωσσική ποικιλομορφία σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη. Uh, also, as a research discipline, Λοιπόν, ε, μελετήθηκε εκτενώς από τη δεκαετία του 50 τεχνητή νοημοσύνη. Την τελευταία δεκαετία όμως βλέπουμε ε, μαζική διάδοση τεχνολογίας ε, τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανικά προγράμματα, προσωπικές συσκευές είναι η πιο καυτή τεχνολογία και συζητείται εκτενώ από τους ερευνητέ, αυτού που διαμορφώνουν την πολιτική, αυτού που κινούνται πρακτικά στον τομέα και διάφορε κοινότητε. Είναι μια πραγματικότητα τεχνητή νοημοσύνη. Διαδίδονται νέε εφαρμογέ, σχεδόν καθημερινά. Και επηρεάζεται και η συναισθηματική κατάσταση από την τεχνητή νοημοσύνη. αλλά βέβαια έχει και αποτέλεσμα να χάνονται θέσει εργασίας. Γιατί γίνονται αυτά. Προσπαθούμε να δώσουμε ανθρωπόμορφη εικόνα στα ρομπότ και στις συσκευές. Η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ θολή και γενική. συγκρίνεται με την ανθρώπινη δυνατότητα για οπτική αντίληψη, ηχητική αντίληψη, μετάφραση γλωσσών, μηχανήματα που μπορούν να μιμηθούν την ανθρώπινη ευφυΐα. Τα μηχανήματα που μπορούν να το κάνουν αυτό θεωρούνται σαν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ομάδα ε, ε, ε εμπειρογνωμόνων δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Τεχνητή Νοημοσύνη και καθορίζει τα συστήματα που δείχνουν έξυπνη συμπεριφορά ότι έχουν τεχνητή νοημοσύνη όταν αναλύουν το περιβάλλον και αναλάβουν κάποια δράση ε, σχετικά αυτόνομα για να πετύχουν συγκεκριμένου στόχου. Δηλαδή, αυτέ οι δράσει δεν είναι προκαθορισμένε ούτε προγραμματισμένε. Τα συστήματα δυναμικά προσαρμόζονται στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Να αναφέρω ότι ο Ευρωπαϊκό Δημιουργικό Τομέα και κυρίω οι συγγραφεί είχαν βασικό ρόλο στη διαμόρφωση του πλαισίου για τεχνητή νοημοσύνη. Το 1943 Η κόρη του Λόρδου Βίρονα δημιούργησε αυτό που θεωρείται ίσως το πρώτο, τον πρώτο αλγόριθμο. Και 80 χρόνια αργότερα ο όρος ρομπότ μάλλον το 1923 δημιουργήθηκε από τον Κάτο Τσάπεκ, ε, τσέχο συγγραφέα, ο Κάρελ Τσάπεκ, στο έργο του RUR. από το ραμπότα που σημαίνει το στα τσεχικά. Όπως ανέφερα, τις τελευταίες δεκαετίες η τεχνητή νοημοσύνη έτυχε μεγάλης προσοχής. Και σήμερα τα περισσότερα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται επί αλγορίθμων εκμάθησης που χρησιμοποιούν τα μηχανήματα. Είναι ευρωνικά δίκτυα όπως αποκαλούνται. Δεν θέλω που προσπαθούν να βγάλουν κάποια μοντέλα γνώσης από δεδομένα. Τα δεδομένα είναι πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη τεχνητή νοημοσύνης. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί η κριτική μάζα για να χρησιμοποιήσουμε εφαρμογέ. Και χρειάζεται μεγάλη υπολογιστική ισχύ για επεξεργασία των αλγορίθμων. Πρόσφατα, μόνο τώρα, έχουμε τέτοια υπολογιστική ισχύ χάρη και στην ε, σοφή χρήση των ε, επεξεργαστών ε, επεξεργασίας γραφικών. Τα συστήματα που αναγνωρίζουν εικόνες, να διαγνώσουν ασθένειες, να ζωγραφίσουν καμπύλες, να μεταφράσουν γλώσσες μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Είναι πολύ ισχυρό εργαλείο η τεχνητή νοημοσύνη για να αντιμετωπιστούν διάφορες ανάγκες πιεστικές και οικονομικές και κοινωνικές. Γι' αυτό τι βλέπουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεταμορφωτικό χαρακτήρα και επιφέρει συγκλονιστικές εξελίξεις σε διάφορους τομείς και έχει γίνει ένα νέο σύνορο για ανταγωνιστική γεωπολιτική προσέγγιση. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σε μια παγκόσμια έκθεση αναφέρεται στο γεωπολιτικό ανταγωνισμό της τεχνητής νοημοσύνης και θεωρεί ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τον πλανήτη. Γεωπολιτικά, άμα δούμε τις προσεγγίσεις που ακολουθούν οι διάφορες περιοχές του κόσμου, βλέπουμε ότι οι πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Κίνα η έρευνα γίνεται κυρίως από την κυβέρνηση. Γίνονται και ιδιωτικέ και δημόσιες επενδύσεις για τεχνητή νοημοσύνη στην Κίνα. Και χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη στην Κίνα και τον έλεγχο της κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι πιστή στις πολιτισμικές της προτιμήσεις και στα υψηλά πρότυπα προστασίας κατά κοινωνικών κινδύνων που δημιουργούνται από τη τεχνητή νομοσύνη. Γι' αυτό φιλοδοξία της Ευρώπης είναι να γίνει περιοχή του κόσμου θα ηγηθεί στην τεχνολογία εχμής, στην τεχνητή νοημοσύνη, συμμορφούμενη όμως με κανόνες. Ανταγωνιζόμενοι όμως το παγκόσμιο προσκήνιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχετικώ εκδώσει ανακοίνωση. Εν 2018. Κοιτάξτε το δημιουργικό κλάδο. Συγγραφής, σκηνοθέτες βοηθούν να διαμορφώνουν τη συζήτηση περί τεχνητής νοημοσύνης, θετικά και αρνητικά στοιχεία, ωφέλη και κίνδυνη. Ήδη το 1949 ο George Orwell, στο περίφημο οδήγημά του 1984, αναφέρθηκε στον ολοκληρωτικό έλεγχο του λαού μέσω εφιούς τεχνολογίας. Αυτές οι τεχνολογίες ήδη υπάρχουν. Ο Στίβεν Χόκινς σε μια ομιλία του στη Σύνοδο Κορυφής του 2017 για το διαδίκτυο είπε, αναφερόμενος στους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης, η αύξηση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι το καλύτερο ή το χειρότερο που θα συμβεί ποτέ στην ανθρωπότητα. Και ίσως πρέπει να σταθούμε μια στιγμή και να εστιαστούμε όχι μόνο στην αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά να δούμε και πώς θα μεγιστοποιήσουμε τα κοινωνικά ωφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτήν. Ξανά, πάνω από 50 χρόνια πριν, στο περίφημο, στην περίφημη ταινία 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος, ο, ο Stanley στην Οδύσσια του Διαστήματος περιέγραψε την κατάσταση κατά την οποία τεχνητή νοημοσύνη όπως ο υπολογιστής HAL 9000 γίνεται ανεξέλεγκτος και θέτει σε κίνδυνο ο HAL το πλήρωμα και το διαστημόπλιο. Και υπάρχουν και άλλα δημιουργήματα, διηγήματα, ταινίε πάνω σε αυτό. Σημαντικά όλα αυτά για να πλαισιώσουμε τη συζήτηση όσον αφορά τα ηθικά θέματα όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Απασχόληση. Εξαλείφθη θέση εργασία η τεχνητή νοημοσύνη. Τι πρέπει να κάνουμε για να διαφυλάξουμε την ε, απασχολησιμότητα. Να είναι δίκαιη η τεχνητή νοημοσύνη. Ο πλούτος που παράγεται από τα μηχανήματα και από τις εφαρμογές, πώς θα ε, μοιράζεται ε, ισότιμα η ανθρωπότητα. Θα διαφυλάξει τις ανθρώπινες αξίες με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και πώς θα διορθώσουμε τα λάθη μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και ποιος είναι υπεύθυνο για τυχόν λάθη λοιπά. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου για την τεχνητή νοημοσύνη έχει καθορίσει δεντολογικούς κανόνες. Στον τομέα τέχνης και πολιτισμού έχουμε κανόνες. Σημαντικός τομέας για τη συζήτηση. Διότι είναι ο χώρος έκφρασης της ανθρώπινης διάνοιας Σκέψεις. Συμμετέχουν ενεργά οι δημιουργικοί πολίτες. Πρέπει να καταλάβουμε εκεί η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης τι συνέπειες έχει. Βλέπουμε πολύ δημιουργικές εφαρμογές, όπως στην μόδα, στην βιομηχανία, στην παραγωγή μουσικής μέσω τεχνητής νοημοσύνης, για την παιδεία. Τα chatbots βοηθούν τα παιδιά να μάθουν νέες γλώσσες. Και γίνανε πειράματα στη Λετωνία μπορεί να φτιάξει και ποίηματα. Όπως ο, ο Ρα, μάθαμε, προσαρμόζει τεχνητή νοημοσύνη σε εφημισμένους ποιητέ, όπως το Ράινις. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την πολιτισμική διάσταση. Πρέπει να ενταχθεί στην παιδεία αυτή η πτυχή, να δούμε τι κινδύνους μπορούμε να αποφύγουμε όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη στα πλαίσια στρατηγική σχετική στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε εθνικό επίπεδο. έχουμε φορείς που εκπροσωπούν τους μεγάλους, μεγάλες επιχειρήσεις και τους ακαδημαϊκούς που επεξεργάζονται πολλά στοιχεία. Όλοι αυτοί επεξεργάζονται τις συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα για τεχνητή νοημοσύνη, σχετικές προτάσεις, πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, δεξιότητες, γνώση, παιδεία, όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση στρατηγικής πρότασης που ετοιμάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει και την πολυγλωσία στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έχουμε 24 επίσημες γλώσσες και 60 άλλες γλώσσες που ομιλούνται ευραίως σαν μικρές περιφερειακές γλώσσες και γλώσσες μειονοτήτων. Η πολυγλωσία είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας και ευρωπαϊκή αξία. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα διαφυλάξει και θα τροφοδοτήσει αυτή την πολυγλωσία. Θα πρέπει να είναι πολύγλωση η ευρωπαϊκή τεχνητή νοημοσύνη. Ιδιαίτερα σημαντικό αυτό για μικρότερε γλώσσε, όπω είναι η μητρική μου γλώσσα, τα λετωνικά. Γι' αυτό η κοινότητα των ερευνητών και αυτών που αναπτύσσουν τεχνολογίε για τι γλώσσε, προτείνουν ολιστική τεχνολογία για τις γλώσσες και πλατφόρμα και να ετοιμαστούν κοινότητε ερευνητών και εταιριών για να προωθηθούν όλε οι ευρωπαϊκέ γλώσσε, όλε οι εφαρμογέ τεχνητή νοημοσύνη. Όλοι οι Ευρωπαίοι έτσι θα ωφεληθούν από την ανάπτυξη τεχνητή νοημοσύνη στη γλώσσα του. Ελπίζω αυτέ, μάλλον είναι διαθέσιμε αυτέ οι διαφάνειε για να δείτε περισσότερε λεπτομέρειε που σα παρουσίασα αργότερα. Αυτά και σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για αυτή την γενικότερη επισκόπηση που μας κάνατε. Τώρα η κυρία Ματαζόσκη Φίλιπς έχει το λόγο. Έχετε 10 λεπτά κι εσείς ε, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θα σας δώσω κάποια στοιχεία ε, σχετικά με το βλέσιο της παρουσίασής μου. Η Ουγγρική κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα της ε, ψηφιακής επιτυχίας και μέσα από αυτό δημιουργήθηκε η Συμμαχία για την Τεχνητή Νοημοσύνη τον Οκτώβριο του 2018. Υπάρχουν 74 ιδρυτικά μέλη που είναι εκπρόσωποι από διάφορους τομείς, ε, από τον ακαδημαϊκό τομέα, τις δημόσιες υπηρεσίες, ε, τις επαγγελματικές οργανώσεις λοιπά. Επίσης, ε, η συμμαχία αυτή είναι ανοιχτή στα νέα μέλη. Σήμερα έχουμε 235 μέλη οργανισμούς. Αυτή ήταν η εικόνα δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2020 και όλοι εργάζονται θελοντικά. Ο στόχος αυτής της συμμαχίας βασικά είναι να προωθήσει την Ουγγαρία στο ευρωπαϊκό προσκήνιο στο, ως προς τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Να γίνει δηλαδή ένα σημείο αναφορά στην παγκόσμια κοινότητα τεχνητής νοημοσύνης. Να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων εταιριών μέσα από εκτεταμένη διάχυση και χρήση των εξελίσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ε, να ε, διευκολύνει την συμμετοχή των startup και των μικρομεσαίων στις δραστηριότητες ε, τεχνητή νοημοσύνης μέσα από εταιρικέ σχέσεις και να εμπλακεί ενεργά η κυβέρνηση στο τοπικό οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιώντας ε, διάφορους ε, τρόπους ε, για να έχει πρόσβαση σε αυτό. Οι βασικοί σηματοδότες αυτής της συμμαχίας είναι οι εξής. Ξεκινήσαμε στις 9 Οκτωβρίου του 2018 και στο πρώτο ήμιση του 2019 ξεκινήσαμε την ενεργό μας δράση. Φτιάξαμε ένα τοπικό ε, website ε, για την τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, ε, έχουμε δημιουργήσει ομάδες εργασίας και ανακοινώθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 2019 το σχέδιο δράσης για την τεχνητή νοημοσύνη από τον Υπουργό. Έγινε λοιπόν το πρώτο βήμα και συντάχθηκε η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η αναμενόμενη ημερομηνία για την οριστικοποίηση της στρατηγικής είναι Φλεβάρης-Μάρτης του 2020. Έχουμε έξι ομάδες εργασίας στη, στη συμμαχία μας, στο συνασπισμό μας. Βλέπετε τα διάφορα θέματα που περιλαμβάνονται στους τομείς επικέντρωσης. Έχουμε εφαρμογές και ανάπτυξη της αγοράς, τεχνολογία και ασφάλεια, βιομηχανία δεδομένων, ε, διεθνείς ε, σχέσεις, ε, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, ρυθμιστικά και ηθικά πλαίσια. Δεοντολογικά πλαίσια. Εγώ ήμουνα επικεφαλής στο project για την εκπαίδευση. Όπως βλέπετε όμως υπάρχουν διάφορα project σε αυτή την συμμαχία, σε αυτό το συνασπισμό. Έχουμε εδώ στην εικόνα μας συγκεκριμένα αναφορά στα project για την εκπαίδευση. Για παράδειγμα, δημιουργία και λειτουργία μιας Ακαδημίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Ένα πανεπιστήμιο στο οποίο μπορεί κανείς να μπει, όποιος και αν είναι, και να ακούσει και να μάθει για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεύτερον, μαζική εκπαίδευση σε σχέση με την ζήτηση στην αγορά εργασίας. Ε, ε, αυτό ε, ήταν κάτι του οποίου εγώ ηγήθηκα. Έχουμε τα περιφερειακά ε, hub, τους κόμβους δηλαδή ε, καινοτομίας και γενικά ένα περιβάλλον ε, έξυπνο για να προωθηθεί η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ο σκοπός αυτού του project, του εκπαιδευτικού project, είναι να έχει μία ευθυγραμμισμένη πρόταση προς την κυβέρνηση και προς τον τομέα της εκπαίδευσης και τον ακαδημαϊκό τομέα. Οι βασικοί στόχοι περιλαμβάνονται σε μια πρόταση. Εκεί ε, διευκρινίζουμε και αξιολογούμε τις προκλήσεις που θέτει η τεχνητή νοημοσύνη στην αγορά εργασίας. Αντιδρούμε στις προκλήσεις αυτές με ένα εφαρμόσιμο εκπαιδευτικό σχέδιο. Ταυτοποιούμε και προτείνουμε ένα ξεκάθαρο κατάλογο αρμοδιοτήτων, ειδικά ε, όσον αφορά στη δημόσια εκπαίδευση και στο σύστημα επαγγελματική κατάρτισης, στην νότατη εκπαίδευση, την εκπαίδευση των ενηλίκων και στην περαιτέρω εξειδίκευση. Επίσης, έχουμε διάφορες μορφές εκπαιδευτικές, διαπίστευσης και ένα σύστημα πιστοτικών μονάδων για τη διαλειτουργικότητα. Επίσης, θέλουμε η εκπαίδευση στην τεχνητή νοημοσύνη να επεκταθεί σε όλους και όχι μόνο σε όσους ε, ασχολούνται αποκλειστικά με τον τομέα της πληροφορικής και είναι ακαδημαϊκοί. Να. Οι προκλήσεις στον τομέα της αγοράς εργασίας είναι οι εξής. Αν ε, ε, δείτε ότι στην Ουγγαρία έχουμε περίπου 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, οι 922.000 θέσεις εργασίας ή αριθμός εργαζομένων μπορεί να έχουν επιπτώσεις μέχρι τα τέλη του 2030. Αυτές οι επιπτώσεις, σύμφωνα με τη μελέτη που σας παρουσιάζω, θα ε, πραγματοθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Αυτή η τάση δεν θα σταματήσει. Έτσι όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Επίσης αναγνωρίζουμε ότι θα υπάρξει μια αλλαγή στο περιεχόμενο των θέσεων εργασίας, θα υπάρχουν θέσεις εργασίας που ακόμα δεν γνωρίζουμε. Αυτό το εκατομμύριο άτομα είναι 25% του συνόλου της αγοράς εργασίας. Σε σχέση με αυτό λοιπόν προτείνουμε ένα εκπαιδευτικό επίπεδο που θα περιλαμβάνει όλους όσοι είναι ήδη στο εκπαιδευτικό σύστημα ή θα μπουν στο σύστημα μέχρι το 2030. Προτείναμε λοιπόν αυτή τη διαφοροποιημένη λύση σε εκπαιδευτικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα επίπεδα τυπικής εκπαίδευσης ε, στην Ουγγαρία. Το project περιλαμβάνει διάφορες προτάσεις. Για παράδειγμα, μία για την ε, επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επανεκπαίδευση για τους ε, εργαζόμενου που ενδεχομένω να πληγούν, ε, μια διαφοροποιημένη εκπαίδευση στον τομέα τη τεχνητή νοημοσύνη για του φοιτητέ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο δημόσιο και ιδιωτικό σύστημα εκπαίδευση, μια πρόταση να συναντηθούμε με τις επιχειρήσεις και τον τομέα της βιομηχανίας και να δούμε ποιες είναι οι ε, προσδοκίες τους και να τις εκπληρώσουμε. Ε, πρόταση για μια πιθανή μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματική εκπαίδευσης και κατάρτισης, πρόταση για τη συμπερίληψη της τεχνητής νοημοσύνης και ε, των τεχνολογιών της πληροφορίας στην ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, προτείνουμε να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των διδασκότων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ή ε, πληροφορικής παύλα τεχνητής νοημοσύνης ε, στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. Επίσης, ε, ζητούμε τη δημιουργία μιας συνεργατικής και υποστηρικτικής δομής, ενός περιβάλλοντος δηλαδή, με συντονισμένες δράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και της βιομηχανίας, καθώς και του εκπαιδευτικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο πλαίσιο και την προσαρμογή στις ανάγκες του μέλλοντος. Ε, όλα αυτά σε επίπεδο τεχνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό κτλ. Τα αποτελέσματα τώρα και οι επιπτώσεις του project. <clears throat> Υπάρχει δυνατότητα για τη δημιουργία και αντικατάσταση των ε, εξειδικευμένων εργατών σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ε, δίνουμε επίσης να προβλέπονται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας που αλλάζει πριν από την τελική εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο θα αυξηθεί η απασχόληση και θα μειωθεί η αναμενόμενη ανεργία. Επίσης, θέλουμε να πάμε την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης πέρα από την εκπαίδευση στην απλή πληροφορική. Επίσης, θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στις εφαρμοσμένε βιομηχανίες να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και την δυνατότητα στι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά του. Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας. Παρακαλώ, ποιος έχει ερωτήσεις. Thank you, Madam Chair, for the floor. Uh, I would like to thank both. Ο κύριος Κόχουτ. Ευχαριστώ του ομιλητέ για τι ενδιαφέρουσε απόψει που περιέγραψαν. Έχω μια ερώτηση όσον αφορά το μεταβαλλόμενο ρόλο του δασκάλου, ανθρώπου δασκάλου, στη διαδικασία εκμάθηση. Όταν χρησιμοποιεί τεχνολογίε τεχνητή νοημοσύνη, σε ποια κατεύθυνση πιστεύετε ότι θα γίνουν οι αλλαγέ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συλλέξουμε κάποιε ερωτήσει ούτω ώστε μετά να απαντήσουν οι δύο ειδικοί του πάνελ. Μιχαήλα Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Η παρουσίαση του Ουγγρικού προγράμματος ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Η ανησυχία για τις απώλειες θέσεων εργασίας και για την αλλαγή στα προσόντα και τις δεξιότητες είναι κάτι που πλησιάζει. Ήδη είναι μια πραγματικότητα και φοβάμαι ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών δεν ανταποκρίνονται αρκετά γρήγορα στις αλλαγές αυτές. Ε, στις παρουσιάσεις σας αναφερθήκατε στους βασικούς πυλώνες των στρατηγικών των κρατών μελών όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν υπήρξατε πολύ σαφείς, εξού και ερώτησή μου. Σκοπεύετε να επενδύσετε σε τεχνολογίες, θα αλλάξετε την εκπαίδευση των διδασκάλων, θέλετε να επεκταθούν τα μαθήματα για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, διότι οι πληροφορίες που δώσατε δεν ήταν τόσο συγκεκριμένες πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε την κυρία Σόντροβα, Ανδρέα από uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω ουγγρικά, λέει η κυρία Μπότσκορ. Διότι έχω και κάποια θέματα να θέσω προς τον Ούγγρο συνάδελφο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω ότι η καινοτομία και οι τεχνολογικές εξελίξεις και έρευνα είναι βασικές προτεραιότητες για την Ουγγαρία. Έχουμε ένα ξεχωριστό Υπουργείο αρμόδιο για αυτά τα θέματα, οπότε αποτελεί ο τομέας προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Είναι ένας τομέας, όπως έλεγα, που αποτελεί προτεραιότητα. Η ερώτησή μου τώρα. Μιλήσατε για αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο έχετε συμμετάσχει. Ποιες κοινωνικές ομάδες ήταν ο στόχος σας. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος. Ποιες κοινωνικές ομάδες. Ποιοι τομείς καλύπτονται. Είναι σημαντικό πιστεύω να δούμε πόσο μεγάλη είναι η κάλυψη αυτού του προγράμματος όσον αφορά την κοινωνία. Ευχαριστώ. Ναι, σε αυτό το σημείο θα σας δώσω την δυνατότητα να απαντήσετε, να κάνουμε μια παύση στις ερωτήσεις και μετά θα συνεχίσουμε. Καταρχάς, αν με επιτρέπετε, να απαντήσω στην κυρία Μπότσκορ Ποιες κοινωνικές ομάδες καλύπτονται. Στην πράξη όλοι. Άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε κανονικές συνθήκες και άνθρωποι σε εξαιρετικά μειονεκτικές θέσεις. Αυτό δεν το ανέφερα στην παρουσίασή μου, αλλά κάναμε μια πρόταση στην κυβέρνηση ε, για ένα ειδικό πρόγραμμα. Χρειάζονται εταίροι βέβαια ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Οι μειονεκτούσες κοινωνικές ομάδες είναι σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Έχουμε κατάρτιση που παρέχεται για δύο εξάμηνα και περισσότερα, για άλλα δύο εξάμηνα μάλλον. Υπάρχει το βασικό, βασική σχολική εκπαίδευση, συν ένα κολέγιο που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές. Επίσης, χρειαζόμαστε απ' την άλλη και μια πολυεθνική εταιρεία ή πολύ ανταγωνιστική εταιρεία που να συμμετάσχει, που θα αναλάβει τον έλεγχο, την παρακολούθηση και που θα παράσχει υποστήριξη στους μειονεκτούντες αυτούς ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι από μειονεκτούσες ομάδες κοινωνικές μετά από αυτή την κατάρτιση μπορούν να συνεχίσουν τη μελέτη τους, τις μελέτες τους, ε, τις σπουδέ τους σε ανώτερη εκπαίδευση. Χρειαζόμαστε την ειδική κατάρτιση λόγω του συστήματος ε, βαθμολόγιστης. Έχουμε αρκετά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτό το τομέα και είμαστε διαπραγματεύσεις με τα σχολεία. Ε, ποιοι τομεί καλύπτονται? Σχεδόν όλοι οι τομείς, από υγεία, στην παιδεία, τα πάντα, όλοι οι τομείς καλύπτονται αυτό, από αυτό το πρόγραμμα ή επηρεάζονται από το πρόγραμμα, διότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει αντίκτυπο παντού. Και βέβαια η παιδεία και αυτή ε, υπόκειται σε αυτόν τον αντίκτυπο. Και συνεχίζω ε, με αντίστροφη σειρά στις τεθήσεις ερωτήσεις. Η κυρία Σόιντροβα έκανε μια ερώτηση. Αν λησμονήσω μία ερώτηση, υπενθυμίστε το μου παρακαλώ. Η κυρία Σόιντροβα λοιπόν ρώτησε για αυτό το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλη σημασία στην Ουγγαρία. Αν θυμόσαστε τον πίνακα που σας έδειξα, που έδειχνε όλα τα προγράμματα, όλα αυτά ανήκουν στην Εθνική Στρατηγική και το σχέδιο δράσης για την τεχνητή νοημοσύνη επίσης. Όλα αυτά αποτελούν ένα κομμάτι του όλου σχεδιασμού και βέβαια χρειάζονται επενδύσεις. Επενδύσεις σε τεχνολογία, σε πολλούς τομείς, αλλά οι εταίροι βεβαίως θα κάνονται τις επενδύσεις. Είμαι επικεφαλής του προγράμματος για την παιδεία. Επενδύουμε λοιπόν στον τομέα της παιδείας. Ο προλαλής σας συνάδελφος αναφέρθηκε σε κάποιους φόβους, κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την αγορά εργασίας. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να είμαστε προετοιμασμένοι. Είναι καλύτερα να φοβόμαστε λίγο και να προετοιμαστούμε παρά να ευνηδιαστούμε αργότερα γιατί πήγαμε αμέριμνοι και κινηθήκαμε αμέριμνα προς το μέλλον. Η ομάδα εργασία προσπαθεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λύσεις, τη τεχνητή νοημοσύνη. Κινούμαστε σαν υπάρχει ε, ανοιχτό πανεπιστήμιο. Όλοι μπορούν να μάθουν, όσοι δεν συμμετέχουν στην επίσημη εκπαίδευση, στη μαζική εκπαίδευση, όλοι μπορούν να συμμετάσχουν. Χρειαζόμαστε όλη την κοινωνία, πρέπει να προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε όλους σε αυτού του είδους την εκμάθηση. δεν ξέρουμε ποια θα είναι η μορφή του μέλλοντος, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε και για ενδεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Είσαστε ικανοποιημένοι, ελπίζω, με τις απαντήσεις μου. Έτσι. Και μετά, α, είχα και μια τρίτη ερώτηση, αν θυμάμαι σωστά. Ο ρόλος του δασκάλου, με ρωτήσατε, αν θυμάμαι σωστά. Ποιος είναι ο ρόλος του δάσκαλου μέσα σε όλα αυτά. Ο ρόλος των διδασκόντων. Α, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αντικαταστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, διότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι η αξία, η βασική είναι το ανθρώπινο «ον». Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό. Ας χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για καλό σκοπό. Υπάρχει και μια οργάνωση που έχει τον τίτλο «Τεχνητή νοημοσύνη για το καλό». Μπορούμε να μιλήσουμε και για την ηλεκτρονική εκμάθηση στο διαδίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξουμε όλους τους δασκάλους και θα τους αντικαταστήσουμε με την τεχνολογία. Πώς να το θέσω τώρα. Κοιτάξτε, στην παιδεία οι μαθητές ήδη χρησιμοποιούν την ψηφιοποίηση. Οι φοιτητέ στο πανεπιστήμιο είναι σε επαφή με αυτή την τεχνολογία με τους καθηγητές τους και η ηλεκτρονική μάθηση, εκμάθηση έχει και άλλες μορφές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειαζόμαστε διδάσκοντες, διότι ο διδάσκαλος μπορεί να δώσει διαφορετικές απαντήσεις δεν ακολουθεί αποκλειστικά έναν αλγόριθμο δάσκαλος και μπορεί αναπερίπτωση να δώσει παιδεία ανάλογα με την ανάγκη του κάθε φοιτητή μαθητή. Ευχαριστώ. Thank you. σας ευχαριστώ. Έχω και εγώ να σας πω δύο λόγια όσον αφορά το ρόλο του διδάσκοντος. Η τεχνητή νοημοσύνη ε, μπορεί να σχηματίσει και να βελτιώσει τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν οι διδάσκοντες αλλά και οι άνθρωποι γενικότερα. Θέλει να παρέχει ε, κίνητρα, στήριξη στην απόκτηση δεξιοτήτων ε, και να τους κατευθύνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ψηφιακή εποχή. Μιλάμε για την ψηφιακή, ψηφιακό αλφαβητισμό. Θα πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για αλφαβητισμό στην τεχνητή νοημοσύνη για να δείξουμε πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να ε, βοηθήσει και πώς μπορούν οι άνθρωποι να υποφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Ο ρόλος του δάσκαλου, του δάσκαλου είναι σημαντικός, είναι ουσιαστικός, αλλά αλλάζει και επίσης ως δημιουργή νέων πλατφορμών μάθησης που βασίζονται στην ε, τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουμε ας πούμε παραδείγματα στην Λετωνία όπου οι δάσκαλοι συμμετέχουν στην ανάπτυξη ας πούμε ε, ρομπότ ε, ομιλίας για να, που βοηθούν στην εκμάθηση γλωσσών και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε ότι αυτός ο τομέας είναι σε καλύτερη θέση από άλλους ε, γιατί είναι πολύ σπουδαίος ε, και μεγάλος τομέας, η τεχνητή νοημοσύνη στην ουσία αναλαμβάνει ε, κομμάτι της βαρετής ε, και μονότονης δουλειάς. Το δημιουργικό κομμάτι παραμένει για τους ανθρώπους, αλλά είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι πολιτιστικές πτυχές του τομεί ε, της στρατηγικής, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενίσχυση των δεξιοτήτων των καλλιτεχνών, των ε, δημιουργών και των δημιουργικών κλάδων για να καταλάβουν πώς μπορούν καλύτερα να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη και τους, για να δημιουργήσουν νέες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, να υπάρξουν χώροι που μπορούν να, να μοιραστούν στοιχεία και διαφορετικά στοιχεία ώστε να καταλάβουμε πολλές επιτυχές ε, ανάπτυξης ε, από διαφορετική προοπτική. Επίσης, να ενθαρρυνθεί η νέα, νέα αγορά ε, για την τέχνη, γιατί και η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάποιες φορές τέχνη να ενθαρρυνθούν τα πολιτιστικά ιδρύματα να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν ειδικού χώρους και ε, ε, δημιουργίες ε, καλλιτεχνικές που θα δείξουν και θα αναδείξουν το πλούτο του ευρωπαϊκού πολιτισμού με έναν νέο τρόπο. Αυτό σημαίνει όμως στοχευμένες δράσεις και αυτό που κάνουμε είναι στις εθνικές στρατηγικές ε, να, προσπαθήσουμε να στραφούν περισσότερο. Ευχαριστώ. Έχω και εγώ ίδια μια ερώτηση. Αν μπορούσα να έχω μια απάντηση ε, πριν δώσω στην Κομισιόν στον πρώτο γύρο την, τον λόγο, εκτός αν υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τους ευρωβουλευτές. Όχι, δεν βλέπω. Άρα επανέρχομαι στο θέμα της εκπαίδευσης και της δημιουργικότητας. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της ψηφιοποίησης, της ηλεκτρονικής μάρτισης και της τεχνητής νοημοσύνης. Τα νέα αυτά συστήματα εξελίσσονται, επεξεργάζονται μεγάλο αριθμό δεδομένων και γενικά υπάρχει ένα μεγάλο περιεχόμενο σε όλη την Ευρώπη το οποίο μπορεί να συγκεντρωθεί και να δημιουργηθούν νέα προγράμματα σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ε, μαθητή και τις απαιτήσει ε, μέσα από τα πλαίσια της τεχνητής νοημοσύνης. Ε, έτσι λοιπόν είναι δυνατό ε, να έχουμε μια δημιουργική συνεργασία και να υπάρχει ένα μάθημα το οποίο είναι τελείως διαφορετικό, όχι μόνο ένας που διδάσκει, να υπάρχει μια επαφή με το μέσο πολύ διαφορετική. Υπάρχει μια υποστήριξη, ε, να ενισχύει συναισθηματικά, να υπάρχει μια διαρθρωτική αλληλό υποστήριξη και μάθηση, περισσότερα περιεχόμενα, και συγκέντρωση συγκεκριμένων δεδομένων και ενιο ενιών. Λίγο κοιτάζω προς το μέλλον, γιατί πρέπει να σκεφτούμε ε, τα βήματα που θα κάνουμε ώστε να μην μείνουμε πίσω. Το και για τον τομέα της δημιουργικότητας, ήδη σήμερα. Υπάρχει αυτή η νέα δυνατότητα, ας πούμε, το New Rembrandt, ε, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να φτιάχνουμε έργα ε, που μοιάζουν με αυτά συγκεκριμένων δημιουργών. Έτσι, ε, να φτιάχνουμε καινούργια περιεχόμενα. Πόσες νέες δημιουργίες εντός εισαγωγικών μπορούμε να φτιάξουμε με βάση τον Ρέμπραντ ή άλλους ε, παλαιότερους καλλιτέχνες. Είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, είναι κάτι που θα μας δώσει μια καινούργια πραγματικότητα και πραγματικά ποιος είναι ο ρόλος της δημιουργικότητας εδώ, ποιος είναι ο καλλιτέχνης. Αυτά που μαθαίνει κανείς σε μια σχολή καλών τεχνών ε, τελικά δεν έχουν μεγάλη διαφορά από αυτά που μπορεί να κάνει μια μηχανή. Απλώς κάθονται κάτω και βάζουν και συνθέτουν εικόνες με βάση στοιχεία που ήδη υπάρχουν. Και τι είναι ο καλλιτέχνη, ε, παίρνει πράγματα τα οποία ήδη υπάρχουν και τα αλλάζει, τα μετατρέπει και τα συνδυάζει με άλλο τρόπο για να φτιάξει κάτι καινούριο και δημιουργικό. Το, αυτό το κάνει και η τεχνητή νοημοσύνη πια. Πού είναι λοιπόν το σύνορο και το όριο μεταξύ ε, τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινης τέχνης. Yeah, um, Thank σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Να δούμε ε, υπέροχες νέες ευκαιρίες και τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στην απελευθέρωση ε, όλων των δυνατοτήτων των ανθρωπίνων όντων. Διευκολύνει τη δημιουργικότητα, αλλά δεν αντικαθιστά τους ε, ε, ανθρώπους. Ένα παράδειγμα που μπορώ να αναφέρω ως προς αυτό είναι η βιομηχανία μόδας, όπου μία σχεδιάστρια, η Τζέσικα Σμάρτ, για παράδειγμα, συνδύασε διάφορες συσκευές με νέο είδος ε, ειδών μόδας που είναι σχεδιασμένα με καλλιτεχνικό τρόπο ώστε να βοηθήσουν ανθρώπους με, ε, με ε, προβλήματα κινητικά, ανθρώπους που έχουν υποστεί κεφαλικό ε, γιατί ε, τα ρούχα αυτά που χρησιμοποιούσε, ε, που, που έφτιαξε μάλλον, είχαν διάφορους αισθητήρε και βοηθούσαν τους ανθρώπους αυτούς να ξεπεράσουν την αναπηρία τους. Άλλο παράδειγμα είναι η βιομηχανία της μουσικής που υπάρχουν νέες τεχνικές για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί η μηχανή με στοιχεία που βάζουν οι άνθρωποι όπου δεν χρειάζεται κανείς να είναι μουσικός, ούτε να έχει μουσική παιδεία, αλλά μπορεί να κατευθύνει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και να δημιουργήσει ένα προσωπικό ήχο. Η τεχνητή νοημοσύνη αντισταθμίζει την έλλειψη ειδική γνώσης της μουσικής σε αυτή την περίπτωση. Και αυτά είναι απλά κάποια παραδείγματα εάν χρησιμοποιηθεί σωστά η τεχνητή νοημοσύνη ε, ενισχύει τη δημιουργικότητα των ανθρώπων αυτό που είναι σημαντικό να καταλάβουμε ε, και να κάνουμε είναι να χαράξουμε μία γραμμή ανάμεσα στην ε, καλλιτεχνική έκφραση που δημιουργείται μόνο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και της ανθρώπινης δημιουργικότητας που υποβοηθείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα είναι εύκολο. Επίσης, τι είδους ε, πνευματικά δικαιώματα μπορεί να απαιτήσει κανείς για τα δημιουργήματα των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα μιλάμε για αλλαγές στην παιδεία. Σωστά αναφέρεται την ε, εξατομίκευση και την προσωποποίηση της ε, εκπαίδευσης. συστήματα που αναπτύσσονται τώρα βοηθούν ώστε η η εκπαιδευτική ύλη, η διδακτέα ύλη να ε, ε, κατακαιρματιστεί σε μικρά κομμάτια μέσα στα οποία κατευθύνει η τεχνητή νοημοσύνη των μαθητευόμενων, τον μαθητή. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού λοιπόν είναι σημαντική όχι μόνο λόγω της νέας τεχνολογίας αλλά και για τους ε, ειδικού και, και δασκάλους καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργείται από τους ανθρώπους και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί είναι το κλειδί για την δημιουργία συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και τη χρήση τους σε μαζική κλίμακα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχω και εγώ να κάνω κάποια σχόλια που αφορούν ε, το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού. Έχουμε σχεδιάσει και έχουμε κάνει ένα ολόκληρο εκπαιδευτικό ε, πρόγραμμα και είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες του κάθε κλάδου και ε, για να μπορέσουμε να αποφύγουμε αρνητικό αντίκτυπο. Βέβαια υπάρχει κάποιο είδος ε, προσωποποίησης ή ειδίκευσης γιατί μπορείς να διαλέξεις αν θα θέλεις να ακολουθήσεις τον κλάδο των, ε, της επιστήμης των δεδομένων ή κάποια άλλη κατεύθυνση ρομποτική ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να καλύψουμε όλες αυτές τις ανάγκες ε, της βιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ. Κομισιόν. DGR, DG Connect. Ευχαριστώ πολύ από την DG Connect. Ένας στους βασικούς πυλώνες του πακέτου που υιοθετήθηκε σήμερα, το ψηφιακό πακέτο, είναι η τεχνολογία που λειτουργεί για τον άνθρωπο. Όπως υπόθηκε, θέλουμε να καλύψουμε ευρύ φάσμα δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε ανθρώπους που έχουν τις σωστές γνώσεις και δεξιότητες και ξέρουν περί τίνος πρόκειται και ποια δεδομένα χρησιμοποιούνται. Αυτές είναι οι δράσεις που αντικατοπτρίζονται στη Λευκή Βίβλο για τεχνητή νοημοσύνη και σχετική στρατηγική. Αυτός μεταφράζεται σε ανθρώπου που έχουν τις βασικές ψηφιακές γνώσεις για να κατανοήσουν. Ήδη ο εμπειρογνώμων αναφέρθηκε στην, στον αλφαβητισμό όσον αφορά τη τεχνητή νοημοσύνη και αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού χρειάζεται για να μάθει νέου τρόπου εργασία που αλλάζει η εργασία λόγω τεχνητής νοημοσύνης και να προωθήσουμε τα ψηφιακά ταλέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθηθεί καινοτομία και να προωθηθούν και νέε τεχνολογίε προ χρήση. Αυτέ οι δράσει θα βασιστούν στα ήδη τεκτανόμενα, τα ανέφεραν οι ειδικοί. Το σχέδιο δράση για την τεχνητή νοημοσύνη συμφωνήθηκε από τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τέλο του 2018. Συνεργαζόμαστε βάσει αυτού με τα κράτη-μέλη και εφαρμόζουμε ολιστικές εθνικές στατικικές και Ακούσαμε τι γίνεται και στην Ουγγαρία. Συνεργαστήκαμε με τι άλλε υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιπηλωτικών Δράσεων. Μία από αυτέ διερευνά δυνατότητε νέων προγραμμάτων μαθημάτων και νέου βαθμού εφαρμογών τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορου τομεί και διάφορα σχετικά πτυχία βάσει των γνώσεων. Ε, το νέο πρόγραμμα για την ψηφιακή Ευρώπη που προτάθηκε για το 2021-2027 στα πέσει του προπολογισμού έχει ειδικό κονδύλι για την υποστήριξη ανάπτυξη οτήτων τεχνητής νοημοσύνης μαζί με άλλες προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα DGR. Yes. Good afternoon. Um, Καλησπέρα. Σύντομα από την πλευρά μου να πω ότι σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντική αυτή η ακρόαση. Η Γενική Διεύθυνση ΕΑΚ υποστηρίζει τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μέσω τη μεθόδου ανοιχτού συντονισμού σε όλα τα βασικά θέματα παιδείας και κατάρτισης συμπεριλαμβανομένης τεχνητής νοημοσύνης. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς να πω ότι ήδη διοργανώσαμε δραστηριότητες εκμάθησης μοτήμων στην ομάδα εργασίας για τις δεξιότητες στη Λουμπλιάνα πέρσι. Δυόμιση μέρες συζητήσαμε τρία βασικά θέματα. Αναδιόμενες πρακτικές στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για την παιδεία. Δεύτερον, να μοιραστούμε τρέχουσες ε, πρωτοβουλίες και σχέδια κρατών μελών. Και τρίτον, Συμβάλαμε επίση στη συντονισμένο σχέδιο τεχνητή νοημοσύνη που ανέφερε η συνάδελφος από τη Γενική Διεύθυνση Connect. Μετά, να πω και κάτι άλλο. Στη σχέδιο δράση για την ψηφιακή εκπαίδευση που ξεκίνησε τον Ιανουάριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ιανουάριο του 2018, έχουμε συγκεκριμένη δράση, ειδική δράση για την τεχνητή νοημοσύνη στην παιδεία. Πιο συγκεκριμένα έχουμε δύο πρωτότυπα ε, τα οποία αναπτύσσονται. Το ένα αφορά χάρτη δεξιοτήτων που σχετίζει αποκτηθήσει δεξιότητε σε εκπαιδευτικά προγράμματα με τι δεξιότητε που απαιτούνται από συγκεκριμένε θέσει απασχόληση. Και το αποτέλεσμα του πρωτότυπου αυτού είναι ότι βλέπουμε οπτικά τι ειδικά προγράμματα, τι προγράμματα υπάρχουν για συγκεκριμένε απασχολήσει, ε, για συγκεκριμένε θέσει εργασία και δημιουργούμε νέα προγράμματα μαθημάτων. Μετά έχουμε ένα πρωτότυπο για τον αντίκτυπο που έχει τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορου τομεί. Εκεί το ερώτημα είναι τι είδου τεχνητή νοημοσύνη χρειαζόμαστε για να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους σε τομείς της οικονομίας. Ακούσαμε τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει σχεδόν όλους τους τομείς. Τελικό σημείο, βάσει τη ανακοινώσεω τη ευρωπαϊκή επιτροπή με το ψηφιακό πακέτο, όπου εκεί παρουσιάσαμε μια γενική θεώρηση. φέτο τον Ιούνιο θα επικαιροποιήσουμε και θα προτείνουμε νέο σχέδιο για την ψηφιακή εκπαίδευση. Θέλουμε να εμβαθύνουμε τη δουλειά που κάνουμε όσον αφορά ε, τις προβλέψεις, όσον αφορά την εκπαίδευση και την εκμάθηση μέσω βάση δεδομένων. Χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη για καλύτερα αποτελέσματα και θέλουμε να βοηθήσουμε να αυξήσει η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδα παιδεία, να προετοιμαστούν οι πολίτε για να πάρουν αποφάσει που ε, θα ληφθούν και που θα επηρεάζονται όλο και περισσότερο οι πολίτε από αυτή τη τεχνολογία. Ευχαριστώ. Και τώρα α αρχίσουμε το δεύτερο τμήμα τη ακρόαση. Δίνω το λόγο, την Προεδρία, στο συνάδελφο Μπότσκορ για μερικά λεπτά. Πρώτα η Ελενόρα Ροζάτη έχει το λόγο. Ένα δεκάλεπτο έχει το λόγο η Ελεονόρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Τι θέλω να κάνω στο χρόνο που είναι στη διάθεσή μου. Τρία πράγματα. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα όσον αφορά τη δημιουργικότητα μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Δεύτερον, να διαρευνήσουμε το πώς φτάνουμε εκεί και τι εμπόδια ίσως να αντιμετωπιστούν και τελικά πού πάμε από εκεί και πέρα. Τι είδους νομική προστασία είναι διαθέσιμη για αυτά τα δημιουργήματα που δεν έχουν, έχουν ελάχιστα σχεδόν καμία... Ε, είναι καθαρά δημιουργήματα των μηχανών και των ανθρώπων. Ε, μετά τα πνευματικά δικαιώματα. Είναι ευαίσθητο θέμα τα πνευματικά δικαιώματα παραδοσιακά συνδεόταν με τα δημιουργήματα του πνεύματος, ε, τη δημιουργική έκφραση και μουσικές δημιουργίες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αυτό φαίνεται σαν κάτι που θα το έχετε δει. Ίσως να φαίνεται σαν μια ζωγραφιά του Ρέμπραντ όμως δεν το έκανε ο Ρέμπραντ, όχι. Είναι μια ζωγραφιά που την έκανε η τεχνητή νοημοσύνη, Χρησιμοποιώντα δεδομένα 346 εικόνες του Ρέμπραντ βάλαμε μέσα σε δεδομένα, βάλαμε και αλγόριθμο να μάθει το στυλ ζωγραφικής του Ρέμπραντ και μετά δημιουργήθηκε αυτό, τη τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό Μοιάζει συνηθισμένο, μοιάζει αυτό ο άνθρωπο, μοιάζει σαν το έκανε οποιοδήποτε. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα. Δεν το έκανε ανθρώπινο όνο, αλλά μηχάνημα αυτό το πίνακα. Έχουμε άλλα παραδείγματα στη μουσική. Να σας παίξω λίγο. Κάνα δύο βίντεο. πάμε στη μουσική αυτή που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη. Στο στυλ των Beatles. Τα βέβαια, ε, η στίχη δεν είναι τόσο καλή, αλλά η μουσική ψηλοθυμίζει οι Beatles. Λέει ομιλήτρια. Και εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα. είναι ένα τραγούδι. Δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Είναι διαφορετικό από το προηγούμενο κομμάτι, όπου εδώ το εργαλείο βοήθησε τους μουσικούς, η τεχνητή νοημοσύνη. Στο προηγούμενο παράδειγμα, εκπαιδεύτηκε η τεχνητή νοημοσύνη να φτιάξει δικό της κομμάτι. Δύο παραδείγματα που δημιουργούν διαφορετικά ερωτηματικά το κάθε παράδειγμα. Άλλη περίπτωση. να προχωρήσουμε λίγο με τη διαφάνεια. Ένα doodle που έφτιαξε η Google πέρσι για να γιορτάσει τα γενέθλια του Johann Σεμπάστιαν Μπαχ. Αυτή η εικόνα χρησιμοποιεί στους χρήστες να δημιουργήσουν μουσική με τεχνητή νοημοσύνη σε στυλ Μπαχ. Βάζει τη δημιουργικότητά σου και το doodle της Google δημιουργεί κάτι που ίσως να ακούγεται σαν σύνθεση του Μπαχ. Αυτά είναι όλα παραδείγματα. Και είναι εμφανές ότι ναι μένουμε σε αρχικό στάδιο της τεχνητής νοημοσύνης και δεν κάνει τεχνητή νοημοσύνη κάτι από μόνη της, χρειάζεται ακόμα τροφοδοσία κάποια από τον άνθρωπο, τουλάχιστον στην αρχή, αλλά υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει τεχνητή νοημοσύνη που θα δημιουργεί από μόνη τη αυτόνομα, στο εγγύς μέλλον. Νομικά τώρα, πώς φτάνουμε εκεί. Η απάντηση είναι, πρέπει να έχουμε πολλά κείμενα και δεδομένα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να εκπαιδεύσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Ε, εξόριξης, μέθοδοι εξόριξης γνώσεων και διαδικασίες τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά είναι στο επίκεντρο της τεχνητής νοημοσύνης και στο δημιουργικό πλαίσιο. Όπως ξέρετε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα δεδομένα. Υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά και λέει ότι η αξία των δεδομένων έγκυται στη χρήση τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νομοσύνη για δημιουργία. Στην προηγούμενη θητεία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέτησαν νέα οδηγία που θεσπίζει νέε εξαιρέσει πνευματικών δικαιωμάτων όσον αφορά την εξόριξη δεδομένων και τα δεδομένα. Αλλά ίσω συνεχίσουν να εφαρμόζονται νομικοί περιορισμοί και να εμποδίζουν αυτού του είδου εγχειρήματα και από πλευρά δημιουργική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα στο έγγραφό τη, αναφέρθηκε στην ενδεχομένη ανάγκη αναθεώρηση υφισταμένων κανονισμών ε, και νομοθεσία για πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά, εμπορικό απόρριτο, διότι ίσω δημιουργηθούν νομικά εμπόδια για την τεχνητή νοημοσύνη λόγω αυτή τη νομοθεσία. Το ερωτηματικό που απομένει μετά από αυτά είναι πού πάμε από εδώ και πέρα. Από τη στιγμή που θα έχουμε κάτι που δημιούργησε τεχνητή νοημοσύνη. Προστατεύεται το δημιούργημα από πνευματικά δικαιώματα ή άλλα νομικά δικαιώματα ή όχι. Θα έπρεπε. Εδώ έχω μια ζωγραφιά. Και αυτή δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Στο Obvious Art, βλέπετε στην ιστοσελίδα, ένας αλγόριθμος έφτιαξε τη ζωγραφική και υπέγραψε και την ζωγραφιά ο αλγόριθμος. Πολύθηκε σε δημοπρασία της Κρίστη το 2018 του οίκου Κρίστη πάνω από 400.000 δολάρια είπα επολύθη. Έχετε κάτι πολύτιμο, αλλά δεν ξέρουμε εάν ε, έχει προσαρτημένα κάποια νομικά ε, δικαιώματα. Τι ερωτήσεις πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας. Πρώτα απ' όλα, ο νόμος πνευματικών δικαιωμάτων αναγνωρίζει μόνο ανθρώπους δημιουργούς ή ε, μη ανθρώπινους δημιουργούς ή μόνο ανθρώπους προστατεύει. Δεύτερον, αυτά τα έργα είναι αρκετά τίπα για να προστατευτούν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ενώσεω, αυτό που απαιτείται για να υπάρχει πρωτοτυπία είναι ότι το έργο να έχει προσωπικό χαρακτήρα του δημιουργού. Ε, να είναι αποτέλεσμα δημιουργικών επιλογών του δημιουργού. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρουσιάσει προσωπικότητα, δημιουργικότητα και ελευθερία. Θα το καταφέρει ποτέ. Και τελικά, το πιο ενδιαφέρον θέμα, πρακτικά, Ποιο είναι ο ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων για αυτά τα δημιουργήματα, ο ιδιοκτήτη των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν εκπαιδευτή τεχνητή νοημοσύνη, ο ιδιοκτήτη του μηχανήματο ή τη τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργεί το έργο, είναι το μηχάνημα που έχει νομικά δικαιώματα και καλύπτεται από αυτά. Αυτά είναι εκκρεμή ζητήματα και πιθανότατα θα γίνουν και πιο πιεστικά στο μέλλον. Και έρχομαι τώρα στο τελικό σημείο μου. Είναι κατεπήγον θέμα αυτό να αντιμετωπίσουμε το θέμα πνευματικής προστασίας αυτών των δημιουργημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Αν δείτε τις συζητήσεις που κάνουν οι νομικοί για πνευματικά δικαιώματα παντού, σε όλο τον κόσμο, η τεχνητή νοημοσύνη και το νομικό καθεστώς που τη διέπει, ίσως είναι τα πιο ευρέως συζητούμενα θέματα. Είναι κατεπίγουσα ανάγκη για συζήτηση του θέματος. Μάλλον και ναι και όχι. Διότι τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Είδαμε κάποια παραδείγματα δημιουργικότητας τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί υπάρχει κάποιο στοιχείο ανθρώπινης τροφοδοσίας και πειρασμού. Μπορούμε να επιστρέψουμε πάντα και να βρούμε άνθρωπο, η ανθρώπινη ομάδα που δημιούργησε τεχνητή νοημοσύνη και επέτρεψε στην τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει. Στο μέλλον αυτό ίσως να μην ισχύει. Ίσως να έχουμε παραδείγματα τεχνητή νοημοσύνης που μπορεί να συλλέξει από πηγές δεδομένα, να επιλέξει τι να χρησιμοποιήσει και να δημιουργήσει με τον ίδιο τρόπο όπως εμείς όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο σε μια βιβλιοθήκη και μετά ετοιμάζουμε και γράφουμε το δικό μας μυθιστόρημα. Όμως είναι και πιεστικό ερώτημα διότι αλλάζει ε, η πρόοδό μα πολύ γρήγορα. Είναι κάτι προχωράει πολύ γρήγορα, συμβαίνει τώρα και τα επόμενα 5-10 χρόνια θα έχουμε παραδείγματα πλήρου αυτόνομη τεχνητή νοημοσύνη που θα δημιουργεί από μόνη τη ε, με τη δική τη βούληση δημιουργήματα και θα γίνει πιεστικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είδους νομικό καθεστώς είναι το πλέον ενδεδειγμένο για αυτού του είδους τη δημιουργικότητα. Τα πνευματικά δικαιώματα αυτά κάθε αυτά, τουλάχιστον στην υπηρετική Ευρώπη, παραδοσιακά θεωρούνται σαν φυσικό δικαίωμα του δημιουργού. Δημιουργείς κάτι και έχεις φυσικό δικαίωμα να τύχεις προστασίας. Το ίδιο ισχύει η διαλογική ισχύει για την προστασία δημιουργικότητα τεχνητή νοημοσύνη. σω να είναι δύσκολα τα πράγματα, να υπάρχουν προβλήματα με τα πνευματικά δικαιώματα αυτά κάθε αυτά. Στα πνευματικά δικαιώματα υπάρχουν ηθικά δικαιώματα προσαρτημένα. Το, το δικαίωμα να αναφέρεται ο δημιουργό, ε, να μην στρεβλώνεται το έργο κάποιου από κάποιον άλλον. Αυτά είναι πολύ δύσκολα να τεθούν σε ένα πλαίσιο τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει και το θέμα του όρου προστασία. Η τεχνη... Αρκεί για την 70 χρόνια μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη και τη διάρκεια ζωής ε, του δημιουργού ισχύουν τα πνευματικά δικαιώματα. Στην, στην ε, τεχνητή νοημοσύνη, όταν δημιουργείται νέα εκδοχή, λίγη προστασία. Διαφορετικού είδου προστασία πρέπει να ισχύει. Τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργούν προβλήματα και ίσως τελικά το νομικό καθεστώς που θα έπρεπε να δημιουργηθεί για τα πνευματικά δικαιώματα ε, τη τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι sui generis. Θα πρέπει να προστατεύσουμε και να επιβραβεύουμε την επένδυση εκείνων που επέτρεψαν στην, στην τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να δημιουργήσει. Θα πρέπει όμω να λαμβάνονται υπόψη περιστάσει όσον αφορά την προστασία που χορηγείται και να μην είναι ε, απεριόριστα εκτεταμένοι και να εμποδίζονται άλλα μέρη να δημιουργήσουν ε, άλλες τεχνητές νοημοσύνες, άλλα μηχανήματα λόγω υπερβολικής προστασίας. Σας παρουσιάσω και ένα πρώτο παράδειγμα πλήρους αυτόνομης τεχνητής νοημοσύνης, ο Πινόκιο δημιουργ... Ε, ήταν εξήλυνη μαριονέτα και μετά έγινε παιδί στο παραμύθι. Και τώρα φτάσαμε στην εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να γίνει όλο και πιο αυτόνομη και να μοιάζει όσο το δυνατόν πιο πολύ με εμά του ίδιου. Κάτι σαν τον Πινόκιο, με άλλα λόγια. Λοιπόν, εδώ και κλείνω και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή σας. Όχι σοκαριστική, αλλά μας έδωσε έτσι κάτι για να έχουμε να σκεφτούμε. Ωραία. Τώρα δίνω το λόγο στον Κρίστοφ Κρίνκε για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε αυτήν την παρουσίαση σήμερα. Ονομάζομαι Κρίστιαν Κρόνκι και θα σας παρουσιάσω τις δικές μου σκέψεις για το θέμα των νέων προκλήσεων στον τομέα της οπτικοακουστικής. Όπως θα δείτε στο φυλάδιο που σας μίλησα, ε, υπάρχουν ε, κάποιες έννοιες που σχετίζονται με τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και θέλω να δω πόσο σχετικά είναι όλα αυτά με τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν ε, κάποια συστήματα τεχνητής νοημοσύνης όπου χρησιμοποιείται ένας αλγόριθμος με την ευρύτερη ένα σε ειδικού τομείς της τεχνητής νοημοσύνης. Το εισαγόμενα και τα εξερχόμενα στοιχεία ε, θεωρούνται ότι βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη όταν έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό εξερχόμενης πληροφορίας που βγαίνει από την τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτό γίνεται με αυτονομία και με ευθεία. Υπάρχουν δύο τομείς που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Στον τομέα των οπτικοακουστικών αυτοί που παρέχουν περιεχόμενο και αυτοί που μοιράζονται περιεχόμενο ως πλατφόρμες. Θα δούμε ακριβώς ε, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτών και αυτών που χρησιμοποιούν ενεργά τις πλατφόρμες. Οι παροχή ε, περιεχομένου έχουν μια σειρά πια επιλογών για τη σύνθεση περιεχομένου, όπως το Deep fake που μόλις πριν μας παρουσιάσατε αλλά και θα υπάρχει και μια παρουσίαση μετά επίσης δεν υπάρχει ευφυής, marketing του περιεχομένου ή της δημιουργίας τουλάχιστον ως τώρα. Οι χρήστες ε, ε, αντιμετωπίζονται βάσει των ειδικών προτιμήσεών τους και γενικά με αυτές τις πλατφόρμες ε, Έχουμε λογαριασμούς ε, που δημιουργούν συγκεκριμένα ε, θέματα και περνάνε πληροφορίες με βάση τις τάσεις. Όλα αυτά γίνονται με τέτοιο τρόπο που να φαίνεται ότι η πατρότητα είναι, ανήκει σε κάποιον άνθρωπο για να υπάρχει μια ισότητα στην επικοινωνία. Μιλάμε για τον εξανθρωπισμό της επικοινωνίας ε, μέσα από μηχανές και υπάρχουν και αυτόματοι λογαριασμοί και το FES marketing που μπορούν να δημιουργήσουν την εντύπωση μεγάλου αριθμού χρηστών ε, να μοιράζεται κάποιες ε, πληροφορίες. Είναι σαν μια γνώμη που την ασπάζονται πολύ. Αυτοί που μοιράζονται βίντεο το κάνουν για διαφορετικό λόγο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης πρώτον για να ελέγξουν το περιεχόμενο, να μην υπάρχει παραβίωση της εφαρμοστής νομοθεσίας και για άλλα τέτοια αριθμιστικά ζητήματα. Επίσης, χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για έξυπνο έλεγχο της πρόσβασης της πληροφορίες από μεμονωμένους χρήστες, ε, ας πούμε, για την ε, προσωποποίηση, ειδικά για εμπορικούς σκοπούς. Τέλος, ε, για τη ρύθμιση των υπηρεσιών, ε, των οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Μπορούμε να έχουμε δύο είδη ρύθμισης, προστατευτική ε, ρύθμιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που στην ουσία μας προστατεύει από παραπληροφόρηση ή μη αρμόζουσα πληροφόρηση και δεύτερον που μας βοηθά να αποφύγουμε ένα ανεπιθύμηθο το ή παράνομο περιεχόμενο. Οι χρήστες υπηρεσιών μέσω μαζικής ενημέρωσης ε, εμπιστεύονται περισσότερο το περιεχόμενο που κάποιος ε, συγγράφει παρά αυτό που έχει εμπορική στόχευση. Γιατί στην ουσία είναι πιο αντικειμενικό και δεν έχει την υποκειμενική διάσταση των εμπορικών συμφερόντων. Με αυτόν τον τρόπο, όταν χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί κανείς ε, να πάρει μια απόσταση από το, την εμπορική διάσταση. Έτσι λοιπόν, στα ΜΜΕ δημιουργείται αυτή η ιδέα της προστασίας των καταναλωτών. Τα ατομικά δικαιώματα, δηλαδή η ελεύθερη γνώμη, η ελεύθερη βούληση, στην ουσία προστατεύονται και ε, υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην επικοινωνία που δημιουργείται μέσω, από, μέσω ανθρώπων. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες που τελικά παρουσιάζονται ως ανθρώπινες, ενώ είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που θα πρέπει να πληρούν αυτοί που δημιουργούν περιεχόμενο και το επικοινωνούν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Στην παράγραφο 18 της ε, νέας συνθήκης ε, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη Γερμανία λέει ε, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να δημιουργούνται αυτόματα περιεχόμενα μέσα από τους υπολογιστές. Επίσης, υπάρχει μια προστασία από το ανεπιθύμητο και, μη, και ανάρμοστο περιεχόμενο που περνάει μέσα από τις πλατφόρμες με ή χωρίς την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η διαθεσιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης μας δείχνει ότι στο μέλλον οι πλατφόρμες που μεταδίδουν βίντεο θα πρέπει να είναι σε θέση να φιλτράρουν το περιεχόμενο. Έτσι ώστε να βγάζουν από τη ροή π.χ. τη βία ή την πορνογραφία μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό με φέρνει στο τελευταίο σημείο μου ως προς την κοινωνική σημασία στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και την ευρία αντίκτυπο. Υπάρχει ε, ο νόμος ο οποίος ε, ενδυναμώνει, που βοηθά δηλαδή τους παραγωγούς να έχουν ένα επαρκές επίπεδο ποικιλομορφίας απόψεων. Υπάρχουν κάποια συστήματα φιλτραρίσματος, τα οποία επηρεάζουν και το άτομα και το κοινό γενικότερα. Υπάρχει αυτό το filter bubble ή το echo chamber ως φαινόμενα και τα δύο φαινόμενα έχουν πολύ σοβαρό αντίκτυπο στην διαμόρφωση της κοινή γνώμης. Και υπάρχει η πρόταση αυτά, αυτή η κίνδυνη του φιλτραρίσματος του έξυπνου περιεχομένου να ε, αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένο τρόπο. Για παράδειγμα, στη συνθήκη που ανέφερα που έχει γίνει στη Γερμανία, αναφέρεται η διαφάνεια και η έλλειψη των διακρίσεων ως κανόνες, ε, μοντέλο, ε, στην τροπολογία της οδηγίας για τα οπτικοακουστικά μέσα. Μεγάλη παροχή πλατφόρμας είναι υποχρεωμένη να αποκαλύπτουν τα βασικά κριτήρια της επιλογής, της ισόρευσης και της παρουσίασης του περιεχομένου και τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούν. Για να διασφαλιστεί η πλιάτα των απόψεων, λέει η συνθήκη, δεν πρέπει τίποτα να εμποδίζεται ή να επιτρέπεται χωρίς μία αντικειμενική αξιολόγηση του δημοσιογραφικά επεξεργασμένου περιεχομένου. Υπάρχει επίσης ένας ορισμός των κριτηρίων βάσει των οποίων ε, συγκεντρώνεται, επιλέγεται και παρουσιάζεται το περιεχόμενο. Όμως, λόγω της βασί... βαρύτητας της παρεμβολής δεν υπάρχει νούμερους κλάουζους, ούτε για τους παροχής πλατφόρμας, ούτε για το κοινό. Αυτά θα πρέπει να τα σκεφτούμε ε, μέσα στα πλαίσια της νέας νομοθεσίας. Αυτά είχα να πω μέχρι τώρα και περιμένω τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ξεκινάμε το γύρο των ερωτήσεων. Υπάρχει κάποιος που θέλει να ζητήσει το λόγο? Πέτρα Η Πέτρα Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα καταλαβαίνετε βέβαια. Σκέφτομαι την Ζαμπίνε Φεράνουν που και αυτή μετά από τόσες ε, δύσκολες διαπραγματεύσεις κατάφερε να φέρει πέρα στην οδηγία και τώρα πάλι μιλάμε για την αλλαγή. Τέλος πάντων, σε δύο-τρία χρόνια πάλι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα. Σας ευχαριστούμε κύριε και αναφέρατε το νούμερο κλάουσους. Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε τι εννοείτε, γιατί δεν το κατάλαβα καλά. Ε, haben natürlich auch... Επίσης, μιλήσατε για την υποχρέωση σήμανσης. Ναι, εντάξει. Υπάρχουν διάφορες τέτοιες υποχρεώσεις ε, μέσα στην οδηγία για το Οπτικό Ακουστικά μέσα. Για παράδειγμα, όταν, όσον αφορά στη διαφήμιση. Αυτό το καταλαβαίνω. Όμως, όταν μιλάμε για προληπτικά μέτρα, είμαι λίγο επιφυλακτική. Και όταν μιλάμε για το προφιλτράρισμα του περιεχομένου, δεν με ενδιαφέρει αν αυτά τα περιεχόμενα τα φιλτράρει τεχνητή νοημοσύνη ή ένας άνθρωπος. Αυτό δεν με ενδιαφέρει, γιατί υπάρχει επίπτωση σε θεμελιώδεις ελευθερίες οι οποίες ε, ε, υπάρχει μια επιπτώση τεράστια. και μιλάτε για output και input responsibility. Ευθύνη για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πληροφορίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Τελικά το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε πάντα. Πρώτον, ο περιορισμός της επικοινωνίας. Ο περιορισμός της διαθεσιμότητας περιεχομένου για τους άλλους. Για μένα το ίδιο ακούγονται αυτά. Δεν μου είναι ξεκάθαρο τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο διαχωρισμός και κατά πόσο μπορεί να μας βοηθήσει. Sí, Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ συνδέομαι με την ερώτηση τη συναδέλφου για να σας εκφράσω ένα προβληματισμό μας. Όταν μιλάμε για περιεχόμενο, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τηρήσουμε την οδηγία που υπάρχει και που θα ισχύει και στο μέλλον για αφορά το παράνομο περιεχόμενο γιατί υπάρχει αυτή η οδηγία για τα θέματα ασφάλειας ε, και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό έρχεται σε αντίθεση με την άλλη οδηγία που αφορά την πνευματική διοκτησία. Η τεχνολογία της τεχνικής, τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να βοηθήσει αυτού του είδους τον έλεγχο τη ε, της δηλαδή των κανόνων που ορισμένοι εξ αυτών ισχύουν ήδη στην Ένωση. Η ερώτησή μου όμως έχει να κάνει περισσότερο με την προοπτική αυτή που είπατε ε, για την τέχνη και για την πνευματική ιδιοκτησία πώς επηρεάζεται αυτή. Μιλάμε για ε, το, τα ηθικά, διοντολογικά δικαιώματα. Δηλαδή στην ουσία τώρα μιλάω, σκέφτομαι φωναχτά, αλλά θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας γνώμη. Νομίζω πως εν τέλει η ανάδυση της ε, εφαρμοσμένης ε, τεχνητής νοημοσύνης ε, ε, στην καλλιτεχνική δημιουργία μας φέρνει το πολύ βασικό ερώτημα του τι είναι τέχνη. Εγώ προσωπικά δεν ε, ξέρω ακόμα ακριβώς <laughs> τι είναι τέχνη, δεν έχω απάντηση για να δούμε ακριβώς τι απορρέει όμως όταν δώσουμε την απάντηση. Πνευματικά δικαιώματα, ηθικά δικαιώματα, εγώ πιστεύω πως όχι. Ε, από αυτού του είδους τις εφαρμογές εγώ θα το απέκλεια. Πάντως η τέχνη είναι κάτι το πολύ υποκειμενικό από δύο άποψεις αυτό που το εκφράζει, το, το δημιουργικότητα αυτό που το εκφράζει, αλλά και είναι και τελείω τελείως υποκειμενικό σε σχέση με το αυτόν που το εισπράττει. Ε, κάποια πράγματα μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρα γιατί είναι τέχνη και τι όχι. Όμως αν μιλήσουμε για ένα τραγούδι όπως αυτό, μια μουσική μάλλον που ακούσαμε όπως αυτή που μοιάζει με τους Beatles, τα συναισθήματα που μπορεί να μας προκαλέσει μπορεί να είναι παρόμοια με αυτά που θα είχαμε αν ακούγαμε ένα, το original κομμάτι των Beatles που δεν τους έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας οι περισσότεροι από εμά. Είναι λοιπόν αυτό τέχνη από τη στιγμή δηλαδή που μας ε, προκαλεί κάποια υποκειμενική αντίδραση αυτό που δεχόμαστε, αυτό που εισπράττουμε ως μουσική και το ίδιο βέβαια ερώτημα μπορούμε να θέσουμε για όλων των ειδών τις τέχνες ή τις μορφές τέχνης. Ευχαριστώ. Και εγώ έχω μια ερώτηση για αυτό το θέμα. Όσον αφορά το θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, ε, φαίνεται ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει δημιουργεί πάρα πολλά δεδομένα. Όταν έχω ένα New Rembrandt, όλα αυτά τα δεδομένα καταγράφονται, είναι διαθέσιμα για ανάλυση, επεξεργασία και για να χρησιμοποιηθούν ξανά. Και ο Ρέμπραντ έχει πνευματική ε, ιδιοκτησία με βάση το γεγονός ότι η δική του ιδέα ακριβώς χρησιμοποιήθηκε. Εντάξει, αυτός έχει πεθάνει, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει μια σύγκρουση εκεί. Όταν έχουμε μουσική ε, με βάση ενώ, την δουλειά ενός ε, εν ζωή καλλιτέχνη, Ίσως θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται να ρυθμίσουμε μια κατάσταση βάσει της οποίας δημιουργούνται νέα έργα με την θεματική δουλειά κάποιου που ήδη έχει δημιουργήσει κάτι και πώς ακριβώς ε, τα συστήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να περιλαμβάνουν το data mining, την αλίευση δεδομένων και πώς ε, ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντική ε, για να προστατεύεται η πνευματική ιδιοκτησία ειδικά όταν ο ιδιοκτήτης της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν είναι πλέον εν ζωή. Υπάρχουν φίλτρα ενδεχομένως που μπορούν να μας δείξουν το δρόμο το να έχουμε την δημιουργία ε, ενός έργου τεχνητής νοημοσύνης ε, από την δουλειά κάποιου που ε, δεν ζει, αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια σύμφαση γι' αυτό, για να μπορούμε να ξέρουμε τουλάχιστον κατά πόσο υπάρχει έγκριση κανείς να ασχολείται με αυτό το θέμα, να υπάρχει τέλος πάντων συνειδητή ενασχόληση με κάτι που υπάρχει στο ίντερνετ και που ενδεχομένως ας πούμε αν έχω μια ομιλία του Ομπάμα και την περνάω στο δίκτυο χωρίς να ξέρουν οι χρήστες ότι έχει γίνει μια ανάλυση ή όχι, οι δομές, ε, ότι έχουν μπει σε μια ανάλυση. Όλα αυτά πρέπει κάπως να σημαίνονται, να ε, φαίνονται. να έχουν τουλάχιστον την ε, γνώση ότι εδώ κάτι διαφορετικό συμβαίνει. Μια σύντομη επερώτηση, γιατί το ξέχασα. Μιλήσαμε για το, την υποχρέωση διαφάνειας. Ε, με πρώτη ματιά δεν είναι εύκολο κανείς να δει αν κάτι έχει βγει από την τεχνητή νοημοσύνη ή όχι. Εμείς ως πολιτικοί πώς ε, θα διασφαλίσουμε ότι τηρείται αυτή η διαφάνεια είναι ένα θέμα. Μιλάμε για διαφάνεια. Αλλά αν δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, τελικά αν ε, οι ειδικοί της τεχνητής νοημοσύνης και μας λένε ότι ούτε εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε τελικά πώς έχει ε, δημιουργηθεί αυτό. Εμείς ως πολιτικοί πώς θα εκτελέσουμε, πώς θα εφαρμόσουμε μια νομοθεσία η οποία ζητά τον έλεγχο. Σε ερωτήσεις παρακαλώ για να ξεκινήσει ο κύκλο των απαντήσεων και μετά να μας δώσει και η Κομισιόν τη δήλωσή της. Όχι, δεν βλέπω άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Thank you very much uh, for, uh, for your questions. Uh, Ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να πω ότι και στα πραγματικά δικαιώματα που θετήθηκαν στην οδηγία το θέμα φίλτρων στο άρθρο 17. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει μεγάλες συνέπειες. Θα το αφήσω σε εσά το θέμα. Πάω στο άλλο θέμα. Τι είναι τέχνη. Πώς αναγνωρίζουμε τι είναι τέχνη. Δεν ξέρω αν το συναντήσατε πριν από κάνα δίμηνο. Ο Μαρίτσο Κάρτιλαν στο Μαϊάμι έβαλε μια μπανάνα με σελοτέιπ στον ε, τοίχο και ήταν το έργο τέχνης του. Πολύθηκε 120.000 δολάρια είπα. Αυτό τι είναι, τέχνη? Είναι κάτι που ανήκει στην τέχνη, βέβαια καλή ιδέα. Είναι κάτι που αξίζει προστασίας, θεωρούμενο τέχνη, στα πλαίσια της ερώτησής σας. Να πω ότι νομικά τα πράγματα περιπλέκονται συνεχώς. Λόγω νομολογίας του ΔΕΚ και δημιούργησε πολλά προβλήματα το ΔΕΚ, κυρίως στον τομέα του design, όσο στο σχεδιασμό επίπλων έργων ε, μόδας. Πολλά κράτη-μέλη παραδοσιακά είχαν κριτήριο αισθητικής αξίας. Προστατεύεσαι πνευματικό δικαίωμα, διότι έχεις το έργο σου σε μουσείο, οι κριτικοί τέχνης εκτιμούν το έπιπλο που έφτιαξες. Και τώρα το ΔΕΚ τι λέει λέει ότι αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη. Πρέπει να ακολουθείται η προσέγγιση ίδια στα πάντα που διέπονται από τα πνευματικά δικαιώματα. Πρέπει να είναι ένα έργο, κάτι και πρωτότυπο για να προστατεύεται. Το δικαστήριο απαλλάχθηκε από όλα τα κριτήρια αισθητικής αξίας, ε, υποκειμενικότητας, αντικειμενική προσέγγιση συστήνει. Εάν υπήρχε υπόθεση που θα αφορούσε δημιουργικότητα πνευμα... ε, τεχνητής η προσέγγιση θα ήταν ίδια. Κατά πόσο το τελικό έργο που δημιουργήθηκε, το δημιούργημα, είναι κάτι που θα αξίζει προστασίας βάσει της εγενούς πρωτοτυπίας του έργου. Και έρχομαι στο δικό σας ερώτημα. Κατά πόσο κάτι που δημιουργήθηκε στο στυλ κάποιου είναι πράγματι επιλέξιμο η προστασία. Η απάντησή μου είναι απίθανο. Γιατί? Διότι το πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για πνευματικά δικαιώματα απαιτεί κάποιο ψηλό επίπεδο δημιουργικότητα. Πρέπει να φαίνεται η προσωπικότητά σου. Ελεύθερη δημιουργικότητα. Και αν κάνει ένα δημιούργημα στο στυλ κάποιου άλλου, η δημιουργικότητά σου είναι αρκετά περιορισμένη. Διότι προσπαθεί να πλησιάσει το δημιούργημα άλλου όσο μπορεί ποια είναι η τελική κατάληξη. Όσον αφορά τα έργα τη τεχνητής νοημοσύνη, το μεγαλύτερο ερώτημα τώρα είναι κατά πόσο υπάρχει περιθώριο για μη ανθρώπινη δημιουργία στο πνευματικά δικαίωμα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Σε κάποιε περιπτώσει υπάρχει δυνατότητα βάσει δεδομένων, προγράμματα υπολογιστών. Εκεί η νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ενώση αναφέρει ρητά ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να αναγνωρίσουν νομικά πρόσωπα σαν δημιουργού. Αλλά για τη μουσική, την τέχνη, φαίνεται να ισχύει ότι αυτή η ελευθερία δεν υπάρχει. Ίσως να υπάρχει ένα πρόβλημα εξ αρχής όσον αφορά την απέτηση περί δημιουργού και ακόμα και αν υπάρχει περιθώριο να δημιουργηθεί κάτι από μία άνθρωπο, το θέμα της πρωτοτυπίας θα παραμείνει εκρεμές και θα είναι δύσκολο να διατείνεται κάποιος επιτυχώς ότι κάτι δημιουργήθηκε στο στυλ διάσημου δημιουργού ή να ξαναπροτείνεις το δημιούργημα κάποιο άλλο με άλλο τρόπο, δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι αρκετά δημιουργικό που επισύρει προστασία. Αυτά είναι θέματα. Θα κλείσω βασισμένη σε αυτό που είπατε. Τι σκοπό έχει η πνευματική διοκτησία. Να αναφέρω την παράδοση στην πυροτική Ευρώπη, όπου πνευματικό δικαίωμα θεωρείται σαν φυσικό δικαίωμα του δημιουργού, αλλά αν δούμε και παραδόσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ηνωμένε Πολιτείε, το εθνικό δίκτυο, όπου θεωρείται σαν κίνητρο το πνευματικό ε, δικαίωμα που δίνει η χώρα, γιατί ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα είναι χρήσιμη για την κοινωνία. Πρέπει να δώσουμε άρα κίνητρα για την παραγωγή αυτών των έργων, εάν δίνουμε δικαιώματα στη, για τη δημιουργικότητα της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει ανταπόκριση, ανταπόδοση κάποιο που έκανε επένδυση για να γίνει αυτό το έργο. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και ο κίνδυνος αποδυνάμωσης της αξίας του δημιουργικού έργου αυτού καθεαυτού. Ξαφνικά θα υπάρχει μια εισρωή φωτογραφιών Φερρυπίν που δημιουργεί τεχνητή νοημοσύνη που θα ε, υποτιμήσει πάρα πολύ σοβαρά τις ανθρώπινες φωτογραφίες, γιατί ο ρυθμός δημιουργίας θα είναι τέτοιο που παρόλο που η ποιότητα θα είναι καλύτερη από ό,τι ανθρώπου, θα υποτιμήσει το ανθρώπινο έργο. Παραδείγματο χάρη, ε, ήδη κάποιοι τομεί όπω τι φωτογραφίε υποφέρουν τεχνητή νοημοσύνη, διότι υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσει κανεί φωτογραφίε που παράγονται τάχιστα, δεν δημιουργούν νομικά προβλήματα, διότι δημιουργούν αντικείμενα σύνθετα, άρα δεν χρειάζεται την άδεια να χρησιμοποιήσει την εικόνα κάποιου, ούτε να διαπραγματευτεί δικαιώματα. Άρα έχει ένα εργοστάσιο παραγωγής φωτογραφιών, έργων φωτογραφικών παράγονται τάχιστα. Και δεν είναι σαφέ αν προστατεύονται ή όχι αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο είναι προβληματικό. Και απειλούνται κάποιες παραδοσιακοί, κάποιοι παραδοσιακοί δημιουργικοί τομείς. Άλλη μια ερώτηση αν επιτρέπετε, λέει ο προεδρο Μιλήσατε για έργα που είναι παρόμοια ή στο στυλ κάποιου. Τι γίνεται αν η μηχανή έχει άλλο στυλ, δημιουργεί κάτι καινούριο. Έχεις καλλιτέχνες που επηρεάζονται από άλλους δημιουργούς και έχουν αναφορές στα έργα τους και αυτό θεωρείται το δικό τους δημιούργημα τέχνη. Εάν δημιουργήσει κάτι τελείω καινούριο μηχανή θα κάνετε. Κοιτάξτε λέει. Αν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη που δημιουργεί κάτι το οποίο δεν είναι στο στυλ κάποιου αλλά είναι πρωτότυπο τότε ίσως να υπάρχει περιθώριο να πούμε ότι αυτό το ιδιαίτερο συγκεκριμένο έργο είναι επιλέξιμο για προστασία, υποθέτοντας ότι δεχόμαστε ότι ίσως δεν υπήρξε άνθρωπος που είχε κάνει τέτοιο έργο. Το θέμα του δημιουργού, ποιο δημιούργησε κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Στην Ευρώπη και σε άλλες νομολογίες. Παράδειγμα, στη ΣΥΠΑ υπήρξε υπόθεση. Εκδικάστηκε σε δύο επίπεδα. Ε, λοιπόν, δημιούργημα ενός πυθίκου και αν προστατευόταν το δημιούργημα του πυθίκου. Η απάντηση δεν ήταν ικανοποιητική από το δικαστήριο. Είπε ότι ένα ζώο δεν έχει νομική θέση για να μπορεί να διεκδικήσει δικαιώματα. Ήταν μια τεχνικής φύσεως απάντηση που δεν μπήκε στην ουσία των πραγμάτων. Κατά πόσο ο θεωρείται δημιουργός από πλευρά πνευματική διοκτησία. Δόθηκε απάντηση από την Υπηρεσία Πνευματικών Δικαιωμάτων των ΗΠΑ και αναφέρεται σαφώς ότι δεν καταχωρεί το γραφείο ένα έργο που δημιουργήθηκε από ένα ζώο. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι μια ανθρώπινη δημιουργία δεν έχει θέση στα πνευματικά δικαιώματα των ΗΠΑ. Και πιθανότατα η απάντηση να είναι παρόμοια και σε άλλα κάτι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω στην περίπτωση του Πυθίκου που ζωγράφησε κάτι στη ΣΥΠΑ. Χρειάζεται κάποιο προσανατολισμό σε νομοθετικό επίπεδο για αυτέ τι περιπτώσει. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει. Να ξεκινήσω με δύο διευκρινήσει που αφορούν ουσιαστικά θέματα. Τι εννοώ με κριτήρια φιλτραρίσματο ή νούμερο Νομοθεσία που περιγράφει ότι κάποιο περιεχόμενο πρέπει να ευνοείται όσον αφορά την ομαδοποίηση συλλογή περιεχομένου. Εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Πρέπει να τονίζεται, Φερρυπίν. Ή να μπαίνει στα πρώτα δέκα αποτελέσματα μηχανισμού αναζήτησης μιας πλατφόρμας. Διάκριση μεταξύ ροής και κροής. Και ο κανονισμός. Ρύθμιση εκροής. Κανονισμός που αφορά το συμφέρον των χρηστών που επηρεάζονται από την εκροή των πλατφορμών. Κανονισμός και ρύθμιση ροής. Τα συμφέροντα εκείνων που θέλουν να μοιραστούν κάτι μέσω πλατφόρμας. Είναι διάκριση. Κανονισμός ροής εκροής όπως είπατε. Και ρύθμιση. Αυτά πάνε χέρι με χέρι. Παράλληλα. Τώρα, στην ουσία. Ενεργή δίθηση. Ευαίσθητο θέμα. Συζητήθηκε. Διεξοδικά. Στα πλαίσια της οδηγίας για το πνευματικά δικαιώματα. Συζητήθηκε και βάση του κανονισμού για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους παρόχους οπτικοακουστικών υπηρεσιών. Πρέπει να λάβουμε υπόψη δύο πράγματα. Το πρώτο, Η παροχή πλατφορφών και για εκπομπή βίντεο, εκεί είναι που κολλάει η επικοινωνία. Δημιουργείται συμφόρηση στον ψηφιακό κόσμο. Εκεί είναι το κόλλημα. Όλε οι πληροφορίε περνάνε από τα χέρια του. Μα αρέσει, δεν μα αρέσει, έτσι γίνεται. έχουν τις τεχνικές δυνατότητες να εξετάσουν περιεχόμενο, το φιλτράρουν. Το κάνουν ήδη. Δεν είναι ότι δεν το κάνουν. Η νομοθεσία τι πρέπει να καλύψει. Αν θα πρέπει να υποχρεώνονται να χρησιμοποιούν αυτή τη δύναμή τους με κάποιο τρόπο. Για να εξυπηρετήσουν το κοινό συμφέρον. Δεύτερη πτυχή. οι ψηφιακές πλατφόρμες κατακλείζονται από περιεχόμενο. Και μπορεί να μην ενδείκνυται. Μπορεί να παραβιάζει και τα πνευματικά δικαιώματα το περιεχόμενο. Να είναι ακατάλληλο περιεχόμενο. Να προβάλλεται βία, πορνογραφία, τρομοκρατία κλπ. Αν δεν διορθωθεί αυτό, το ψηφιακό σύστημα για το νομικό σύστημα για το ψηφιακό τομέα θα είναι άχρηστο. Χρειάζεται ένα είδος διήθησης. Είναι αναγκαιότης. Δεν είναι τέλεια. Συμφωνώ ότι χρειάζεται μια ισορροπία. Τα δικαιώματα των χρηστών και τα δικαιώματα των πλατφορμών να προωθούν περιεχόμενο καλύπτοντα από τις θεμελιώδεις ελευθερίες περί Μιλάμε για την τέχνη, η ελευθερία στην τέχνη κλπ. Είναι και τα συμφέροντα των χρηστών που καταναλώνουν το περιεχόμενο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ενεργή διήθηση δεν πρέπει να επιβάλλεται για να προστατεύονται συγκεκριμένα συμφέροντα. Πρέπει να βασίζεται στη σοβαρότητα των, συμφερόντων που πλήττονται, επηρεάζονται αυτό το φιλτράρισμα, αυτή η διήθηση. Βάσει συγκεκριμένου περιεχομένου, παρουσίαση βίας κλπ. κλπ. Αυτό δεν αποκλείεται ο έλεγχος και το φιλτράρισμα. Πρέπει να συζητούμε με τι σχετίζεται αυτή η υποχρέωση. Τέλος. Υποχρέωση ετικετοθεσίας ούτως υπήν. Ενημέρωσης για το περιεχόμενο. Όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, θα είναι κρισίμου σημασίας σε μερικά χρόνια οι χρήστες, το κοινό, να γνωρίζει ποιο περιεχόμενο είναι αληθές και ποιο όχι. Είναι υψής της σημασίας να υπάρχει κάτι που θα προβλέψουμε. Ψηφιακό σημάδι, σφραγίδα. Κάποια υποχρέωση αναφοράς πληροφοριών και το περιεχόμενο. Ετικετοθεσία το συμπίν, που θα ενημερώνεται ο χρήστη για το περιεχόμενο. Θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα να αποφασίσουμε το πώς θα καθορίσουμε ποιο περιεχόμενο δημιουργήθηκε μέσω τεχνητής νοημοσύνης και ποιο είναι το εύρος που καλύπτεται από αυτή την υποχρέωση. Γι' αυτό προτείνω να μην ακολουθήσουμε στενό ορισμό περί τεχνητής νοημοσύνης. Ποια είναι η άποψή μου ότι η τεχνητή νοημοσύνη και τα αλγοριθμικά συστήματα δημιουργούν τα ίδια αριθμιστικά ερωτήματα δεν πρέπει να συζητήσουμε τι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Τουλάχιστον όχι σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά το αυτόματα παραγόμενο περιεχόμενο είναι το θέμα. Ότι αυτό πρέπει να σχετίζεται με την υποχρέωση ετικητοθεσίας ενημέρωσης του χρήστη. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι κατά πόσο οι πληροφορίες είναι αληθής ή ψευδής. Ζούμε σε έναν κόσμο όπου ε, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να δούμε τι περιεχόμενο δημιουργήθηκε από μηχάνημα. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο τώρα. Ποιο θέλει να μιλήσει, ορίστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ που διοργανώσατε εδώ την ακρόαση. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες εισηγήσεις τους. Μιλάμε για τη δημιουργική Ευρώπη και τα μέσα και το τι κάνουμε εκεί για το τομέα των οπτικοακουστικών. Εν γέννη, θέλουμε να εστιάσουμε σε μια μεγάλη μελέτη που θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο ήμιση του έτους που είναι μια μελέτη για την τεχνητή νοημοσύνη με εστιασμό στους ε, δημιουργικούς ε, τομείς, ε, ευκαιρίες και προκλήσεις. Υπάρχει και το θέμα της απασχόλησης, το θέμα της πολιτιστικής επικοιλωμορφίας υπάρχει το θέμα της δημιουργίας, ο αντίκτυπος στην δημιουργία. Έχουμε δει εργαλεία που μπορούν να προβλέψουν αν ένα οπτικοακουστικό μέσο θα είναι επιτυχές ή όχι στο σινεμά ή στην τηλεόραση. Ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος αυτού από καλλιτεχνικής άποψης. Θέλουμε να ξεκολουθήσουμε να παράγουμε αυτού του είδους το περιεχόμενο ή θα πρέπει μια, ένα μηχάνημα να αποφασίζει αν αυτό το συγκεκριμένο έργο με το συγκεκριμένο σκηνοθέτη και ηθοποιό θα πάει καλά ή όχι και άρα δεν θα το φτιάξουμε καν. Αυτά όλα είναι πράγματα που πρέπει να τα μελετήσουμε. Κάτι που κάναμε και που λειτουργήσε πολύ σωστά, αλλά και που δημιούργησε και πολλά ζητήματα, ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα, χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε, και ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τον υποτιτλισμό όπου δουλέψαμε Βοηθήσαμε τον πειραματισμό σχεδόν σε πραγματικό χρόνο γίνεται ο υποτιτλισμός που βεβαίως είναι πολύ θετικό γιατί διευκολύνει οι ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε, περιεχόμενο που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να το δουν, αλλά βέβαια υπάρχουν θέματα που όσον αφορά τους μεταφραστές που είπαν ότι ναι, αλλά αυτό δεν είναι καλό σε αυτό το επίπεδο, είναι μόνο ε, κατά 85% σωστή μετάφραση, ακόμα και για ζωντανές αναμεταδόσεις και θα πάρει θέσεις απασχόλησης. Υπάρχει θέμα λοιπόν όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης και το πότε αυτό το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργήσει και ε, με ωφέλιμο τρόπο. Τελευταίος μιλητής για σήμερα είναι ο καθηγητής Κολουβάη από το Μόναχο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε εδώ. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και είναι εντυπωσιακό. one Έχω μία δουλειά. Δύο δουλειές. Πρώτον, είμαι καθηγητής ε, τη σχολή κινηματογράφου. Βοηθώ τους φοιτητέ μου να πραγματώσουν τις ιδέες τους και η δεύτερη δουλειά μου είναι στην ε, βιομηχανία του κινηματογράφου και ε, του animation. Και συνεχώς ε, κάνω κάτι ψεύτικο, φτιάχνω δηλαδή εικόνες που δεν είναι πραγματικές, που δεν υπάρχουν. Αν θυμάστε, ως παιδιά, Είδαμε κάποιες ταινίες, ε, κινούμενα σχέδια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, στον κινηματογράφο να υπάρχει μια ευθύνη. Αυτό λέω στους φοιτητές μου όταν δημιουργούν εικόνες και ιστορίες με αυτές, με τα συναισθήματα που δημιουργούν, κάνουν αξέχαστες τις ιστορίες αυτές και έχουν μια ευθύνη. Μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο στη σημερινή εποχή οι influencers, αυτοί που επηρεάζουν δηλαδή, είναι νέα δουλειά. Ήρθα λοιπόν να σας μιλήσω για το deepfake. Τι είναι αυτό. Να σας πω ότι έχω κάνει 15 ταινίες Marvel. Έχετε δει στη ζωή σας μια τέτοια ταινία, είμαι σίγουρος. Όλοι σας. Τι είναι το deep fake. Υπάρχει μια τεχνική πίσω από αυτό όλο και περισσότερο οι υπολογιστές είναι σε θέση να δουν, να ακούσουν και να μιλήσουν. Το ξέρουμε αυτό από την καθημερινή μας ζωή. Έχουμε τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, που δεν τα έχουμε ακόμα, αλλά ξέρουμε ότι έρχονται. Και όλοι χρησιμοποιούμε τα smartphones. Smartphone, έξυπνο τηλέφωνο. Από μόνο του η λέξη μας δείχνει ότι υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη. Και αν θέλεις να βρεις μια φωτογραφία που πήρες πριν από πολλά χρόνια και δεν έχεις σημάνει με ένα όνομα τη φωτογραφία, υπάρχει το λογισμικό που σε βρίσκει. Ακόμα και αν η εικόνα δεν είναι καλή, αν δεν υπάρχει καλό focus, ο υπολογιστής μπορεί να αναγνωρίσει, να δει, να κατανοήσει το περιεχόμενο. Μπορεί να ακούσατε τη συζήτηση για τον Irish, The Irishman, την ταινία. Ο Ιρλανδός. Oh, um, uh, Διότι οι ηθοποιοί είχαν ένα ρόλο στον οποίο υποδίωταν κάποιον πολύ νεότερο ο Μάρτιν Σκορσέζε ήθελε να δείξει ε, ότι είναι 30 χρόνια νεότερη. Η εταιρεία που το έκανε αυτό, η εταιρεία George Lucas ILM, χρειάστηκε μήνες ε, για να αναπτύξει εργαστη... Ε, εργαλεία και χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη για να κατανοήσει τα πρόσωπα των ηθοποιών. Να δώσει δηλαδή τα στοιχεία στο software, στο λογισμικό, για να τους φτιάξει πιο νέους για να φτάσουμε σε ένα παράδειγμα που φαίνεται εντάξει, αλλά δεν είναι και τόσο πιστικό ακόμα. Φτιάξανε λοιπόν διάφορες τεχνικές ε, ε, που τις ενσωμάτωσαν στις κάμερες και φτιάξανε αυτά τα πρόσωπα των ηθοποιών για να τους αναδημιουργήσουν και να τους δώσουν διαφορετική μορφή. Τον περασμένο μήνα η YouTube ένας καλλιτέχνης δηλαδή από εκεί πήρε αυτά τα στοιχεία και τα ξαναδημιούργησε όλα με το deepfake σε πολύ καλύτερη ποιότητα. Κοιτάξτε. Στον δικό μου χώρο με τα visual effects, η τεχνητή νοημοσύνη καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο και ε, κάνει τη δουλειά πολλών ανθρώπων που ως τώρα χρειαζόταν. Ακόμα και αν κανείς δεν έχει εκπαιδευτεί σε αυτό το τομέα μπορεί με ευκολία να αλλάξει και να προσωμιώσει πρόσωπα και εικόνες. Να, και σήμερα βλέπουμε τέτοια παραδείγματα πολύ ανησυχητικού περιεχομένου. Για παράδειγμα, αν δώσεις στον υπολογιστή το ερώτημα «Βρες μου ξανθούς πολιτικούς» να, αμέσως θα σου βρει εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες. Και μετά μπορείς να παίξεις με αυτό το περιεχόμενο και ο υπολογιστής κατανοεί την κίνηση. Την υποκριτική, Το τρόπο της, ε, το χρειά της φωνής, το διαφορετικό περιεχόμενο. Μπορεί να πάρει όλα τα περιεχόμενα και να τα αναμίξει. Εδώ είναι μια διαφορετική ανάμιξη. Να, κοιτάξτε αυτό το κλιπ.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 And if this ends up on 22 minutes, remember, they're fake news. Deep. Okay, uh, it's going on for. Um... Συνεχίζει το βίντεο. Αυτό είναι ο Φέικενστάιν. Το περιεχόμενο, ξεκάθαρα, είναι φτιαχτό. Ο τηλεθεατής, ε, ο θεατής αμέσως αναγνωρίζει ότι πρόκειται για deepfake βίντεο, δεν είναι κάτι αληθινό. Μπορεί όμως να μοιάζει με αληθινό το περιεχόμενο και είναι επικίνδυνο. Υπάρχει τώρα ένας αγώνας στο facebook, στο youtube, λογισμικό που προσπαθεί να βρει τα deepfakes. Καθώς αναπτύσσονται λοιπόν τα deep fakes, έτσι αναπτύσσεται και η τεχνολογία που τα ανοιχνεύει. Υπάρχουν χαρακτήρες που είναι τελείως φτιαχτοί, τεχνητοί, έχουν πολλούς followers, δημιουργείται μια ολόκληρη οικονομία, αλλά δεν υπάρχει πίσω από αυτά τίποτα. Το θέμα είναι σε ποιον ανήκει το δικαίωμα ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας για αυτές τις δημιουργίες. Τι είναι αυτό. Είναι ένας ε, εκφωνητής που δεν είναι αληθινός, δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, δεν κάνει απεργία, στην ναι. Κίνα τους χρησιμοποιούν και ο κόσμος νομίζει ότι είναι πραγματική. Επίσης υπάρχει και το revenge porn, δηλαδή η πορνογραφία εκδίκησης, έγκλημα. Κάποιοι που προσπαθούν να καταστρέψουν τη ζωή άλλων με αυτόν τον τρόπο. Και στο στρατό φυσικά υπάρχουν πολλά που γίνονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι εταιρείε λοιπόν προσπαθούν να βρουν τα deep fakes. Αυτές οι εταιρείε που το έχουν αναλάβει πραγματικά έχουν πολλή δουλειά αυτή τον καιρό. Ομολογώ. Εγώ είμαι καλλιτέχνης. Ιστορίες αφηγούμε. Και όλο και περισσότερο χρησιμοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη με τη συζήτηση που είχαμε πριν για το πώς κάνω μια διάλεξη σήμερα, να σας πω ότι δεν είναι εύκολο. Στέκεσαι μπροστά στα παιδιά και τα ξέρουν όλα. Γιατί έχουν το YouTube, βρίσκουν ένα κλιπ στο YouTube και το κάνουν. Πώς μπορώ να τους φέρω κάτι καινούριο. Η θέση μου λοιπόν και ο είναι όλο και περισσότερο η θέση ενός moderator, ενός συντονιστή, ενός ανθρώπου που προσπαθεί να τους κατευθυνεί και να τους δείξει το σωστό και το λάθος. Αυτή είναι η θέση μου. Επίσης, τους δείχνω τις ιδέες. Αυτό είναι κάτι άλλο, η τεχνητή νοημοσύνη. Χρειάζεται ιδέες και οι ιδέες έρχονται από τους ανθρώπους. Αν αρχίσουν οι ιδέες να έρχονται από την τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι πολύ βαρετές νομίζω. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, έχετε ερωτήσεις? Κυρία Άντερσον. Äh, Ευχαριστώ λοιπόν ε, όλους τους εμπειρογνώμενες. Wow, τι να πω. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή. Λοιπόν, είδα ε, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση εκεί μέσα σε εισαγωγικά. Όταν ε, μιλάτε στους φοιτητές σας, μιλάτε περισσότερο ως ε, συντονιστής. Γιατί υπάρχουν τόσες πληροφορίες εκεί έξω που πρέπει να τις διαχειριστούν και τους ε, βοηθάτε να αποφασίσουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα η προσέγγιση σας από τη δική σας πλευρά. Εγώ αυτό το θεωρώ μεγάλο πρόβλημα, το είπε και η κυρία Φερχόγγεν. Ποιος είναι ο ρόλος του διδάσκοντα όταν έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη μπροστά μας. Ναι. Επί της αρχής δεν γίνεται αντικειμενικά πια το μάθημα, διότι υπάρχουν τόσες πληροφορίες, όμως ο μελλοντικός διδάσκων έχει ως καθήκον να αξιολογεί τέτοια πράγματα. Από τη δική του οπτική γωνία. Τεράστια δυνατότητα λοιπόν χειρισμών σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στο επίπεδο των διδασκόντων. Η κυρία Κάμε Φέρντεν ε, δεν είναι εδώ. Ε, το είπε. Μιλάμε για δικαιώματα των πολιτών. Να το πω έτσι ξεκάθαρα, αυτό με φοβίζει. Αυτό που συμβαίνει στις κοινωνίες μας. Τι θα γίνει αν τελικά δεν έχουμε τρόπο να καθοδηγήσουμε τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Όλα αυτά με τρομάζουν. Αυτό θα έλεγα. Μπορώ να απαντήσω. Εκτός μικροφώνου. for your... Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ευχαριστώ για την εμπειρία που μοιραστήκατε μαζί μας. Όπως είπατε, είστε καταρχάς καλλιτέχνης ε, στο animation κινηματογραφιστής μπορεί να γνωρίζετε την κινηματογραφική σχολή της Τσεχίας από όπου έχουν βγει πολύ σημαντικοί δημιουργοί και είστε και καθηγητής. Τι θα λέγατε για την εκπαίδευση στον τομέα του κινηματογράφου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί όπως είπατε πρέπει να αναγνωρίσουμε τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο. Πρέπει να τα διαχωρίσουμε πρέπει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτή τη νέα πραγματικότητα. Τι νομίζετε λοιπόν. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα στην Τσεχία ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια στην εκπαίδευση ε, για τον κινηματογράφο να ζητάμε καθηγητές που να μπορούν να διδάξουν κάτι τέτοιο. Ποια είναι η δική σας εμπειρία. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για αυτή την ε, παρουσίαση που μας κάνατε για το deepfake. Σκεφτόμαστε πολύ τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας στη κριτική, ε, στο κριτικό πνεύμα όσο γίνεται, αλλά αυτό το deepfake είναι μια απειλή που μας ανησυχεί πάρα πολύ και μάλλον στην Ευρώπη ε, έχουμε αργήσει όσον αφορά την συνειδητοποίηση αυτού του νέου κινδύνου και θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε παιδαγωγικές προσπάθειες που να έχουν γίνει για τα παιδιά αλλά και για τους ενήλικες γιατί καταλάβαμε ότι υπάρχει μια καταδίωξη σε τεχνολογικό επίπεδο ανάμεσα σε αυτούς που φτιάχνουν τα deepfake και αυτούς που τα ανοιχνεύουν, αλλά εσείς γνωρίζετε για την ύπαρξη ε, παιδαγωγικών προγραμμάτων που να μπορούν να δώσουν στα παιδιά μας τα εργαλεία για να ε, μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν όταν αυτά είναι κακόβουλα. Γιατί δεν είναι πάντα κακόβουλα, μπορεί να είναι και καλλιτεχνική δημιουργία, όπως είπαμε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κι εγώ μια ερώτηση. Δεν είναι τόσο νομικό όσο διοντολογικό το ζήτημα. Ένα ας πούμε φιλμ με τον James Dean που έχει ήδη πεθάνει και ο οποίος δεν θα θέλει να το παίξει π.χ. Πόσο μακριά μπορεί κανείς να πάει, να χρησιμοποιήσει δηλαδή ένα χαρακτήρα, μια προσωπικότητα. Γνωστοί ηθοποιοί, πολιτικοί, άτομα της δημόσιας ζωής, ε, ανεξάρτητα από το που δραστηριοποιούνται ε, μπορεί να μπουν σε ένα πορνό μέσα ε, το deep fake, για να το πω έτσι ομά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τις θετικές πλευρές. Χρησιμοποιούμε με το θετικό τρόπο τις τεχνολογίες ε, για να φτιάξουμε σκηνές χωρίς να βάλουμε σε εκείνο τη ζωή ανθρώπων όταν είναι επικίνδυνες, αυτά είναι μια χαρά, ε, νόμιμα και καλά. Όμως, αν υπάρχουν ε, παρεκτροπές, τι γίνεται. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα άτομα και την κοινωνία μας από τέτοιες εξέλιξεις. Γιατί όσο μορφωμένο και να είναι κανεί, δεν μπορεί πολλές φορές να αναγνωρίσει αν κάτι είναι πραγματικό ή deep fake. Α πούμε, υπάρχει μια ομιλία του Ομπάμα, ε, στην οποία θα μπορούσε κανεί να βάλει μέσα πράγματα που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, να βάλουν κάτι του βαρουφάκι μέσα. Δεν ξέρω, τέτοια πράγματα. Τέτοια πράγματα. Ε, και δάχτυλο, δείχνουμε με το δάχτυλο όταν έχουμε κάνει κάτι κακό. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες λοιπόν να παρουσιάσει κανείς ε, κάτι ψευδές. Υπάρχουν λοιπόν ηθικά ζητήματα. Και αυτά ως ε, νομοθέτες μπορούμε να το κάνουμε. Να προσπαθήσουμε να βάλουμε σε σωστή τροχιά τις εξελίξεις. Φυσικά ε, όσο γίνεται να δώσουμε τη δυνατότητα στα θετικά να χρησιμοποιηθούν και στα αρνητικά να αποφευχθούν. Ευχαριστώ. Ίσως να είναι πολύ απλό. Τίποτα δεν άλλαξε όμως. Τίποτα δεν άλλαξε. Αν πριν από 100 χρόνια απλά το προσωπούσες κάποιον, το ίδιο πρόβλημα υπήρχε. Το μόνο πρόβλημα εδώ είναι το πιστευτό Τη εικόνας, αυτό που θεωρούμε ότι είναι πραγματικό. Αυτό είναι το μόνο. Αν πας σε μια περιοχή, κάπου, που ποτέ δεν είχαν εμπειρία κάποιου πράγματος και τους το δείξει σαν αληθινό, θα το πιστέψουν, θα θεωρήσουν ότι είναι πραγματικό. Τώρα, το πώς εκπαιδεύουμε τα παιδιά μας ή πώς βρίσκουμε έναν τρόπο να εξηγήσουμε το θέμα στα παιδιά και στους φοιτητές τους λέμε ότι πρέπει να καταλάβουν να μην πιστεύουν τα πάντα πρώτα απ' όλα. Να αμφισβητούν τα πάντα. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Αν δείτε μια ομιλία του Ομπάμα, πρέπει να ξέρετε ότι αυτή είναι μια πηγή. Ποια είναι η πηγή, υπάρχει και άλλη πηγή, υπάρχει άλλη πηγή. Α, διαφορετική, άρα κάτι δεν πάει καλά. Ποιος το έκανε. Αυτό που είπαμε το μικρή εικόνα ήταν ο δόκτωρ Φέικενστάιν, κάποιος που κάνει κομμωδίες με αυτόν τον τρόπο. Το περιεχόμενο που δίνουμε στα παιδιά για να μάθουν από αυτό δεν άλλαξε. Θυμάμαι σχολικά βιβλία. Ήμουν τυχερός να μην γεννηθώ στην Ανατολική Γερμανία, αλλά ξέρω πολλά για την Ανατολική Γερμανία και την επισκέφθηκα την Ανατολική Γερμανία όταν υπήρχε. Αν Δει σχολικό βιβλίο της Ανατολικής Γερμανίας και το συγκρίνει με δυτικό γερμανικό βιβλίο, ήταν παρόμοιο το πρόβλημα, το ίδιο πρόβλημα. Το ξεπεράσαμε αυτό και υπάρχουν πολλέ άλλες χώρες που δεν ξέρουμε ποιο δημοσίευσε τα σχολικά βιβλία, Ποιο παρουσιάζει τη γνώση στα παιδιά. Είναι σωστή η γνώση που παρουσιάζει στα παιδιά. Με τον James Dean, Ήταν πολύ καλές ειδήσει για αυτό τον παραγωγό, χρηματοδότη την ταινία του. Εγώ προέρχομαι από τα κινούμενα σχέδια. Μπορώ να κάνω ποιο χαρακτήρα θέλω. Ο James Dean είναι νεκρός. Το να χρησιμοποιήσει το πρόσωπό του ίσως να είναι ένα θέμα. το να πάρεις κάποια πνευματικά δικαιώματα χρησιμοποιήσει το πρόσωπό του. Ο σκηνοθέτης που ετοιμάζει ένα σενάριο αν τιμωρηθεί που κάνει κάτι λάθος με τον James Dean, αυτός θα τιμωρηθεί. Πορνογραφικό έργο με κάποιον που δεν θέλει να παρουσιάζεται σε πορνό. Αυτό είναι έγκλημα που πρέπει να τιμωρηθεί. Βέβαια. Έτσι ήταν πάντα. Τώρα τι άλλαξε. Ότι πρέπει να καταλάβουμε, να μάθουμε, ότι αν βλέπουμε κάτι, ίσως να μην είναι αληθές. Πριν από 100 χρόνια, ό,τι ήταν στην εφημερίδα τυπωμένο, όλοι θεωρούσαν ότι αυτά είναι η είδηση, η πραγματική είδηση. Είναι τυπωμένο στην εφημερίδα, άρα είναι αληθινό. Τώρα πρέπει να πούμε μισό λεπτό. Μπορεί και να μην είναι αληθινό αυτό που βλέπουμε. Το ίδιο με το ραδιόφωνο, με την τηλεόραση και τώρα με το deepfake. Η νομοθεσία μας είναι καλή για τα πνευματικά δικαιώματα, για να αντιμετωπίσει το θέμα. Δεν θα πρέπει να το φοβόμαστε, διότι ίσως να υπάρξουν κακές αποφάσεις στο μέλλον. Πρέπει να το δούμε πώς είναι. Δημιουργία εικόνας, δημιουργία ηχού, συζητιέται το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων οικονομικών, μέχρι ποιο βαθμό πάνε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει να τα διεκδικήσει ένας ε, ο δημιουργός. Δημιουργήσαμε 50, 15 ταινίες μάλλον Marvel, δημιουργήσαμε περιεχόμενο, έχουμε ένα τμήμα με καλλιτέχνες που εφευρίσκουν. Ο Άριμαν φοράει τη στολή, ο Άιρονμαν Σχεδιάζουν το σχέδιο, παίρνουν την πληρωμή τους αλλά δεν παίρνουν ποτέ μερίδιο των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Marvel έχει τα πνευματικά δικαιώματα και η Disney. Η επιχείρηση πάει καλά, όλα είναι κανονικά, έτσι λειτουργεί. Αλλιώ, αν θες να κάνεις μια ταινία, θα έχεις εκατοντάδες επί εκατοντάδων ε, καλλιτεχνών με τους οποίους πρέπει να μοιραστεί τα κέρδη σου. Είναι αδύνατο να οργανωθεί αυτό και να οργανωθεί και λογιστικά καν. Πώς το βλέπω. Ένας μουσικός συνθέτει μουσική και δίνει ένα κοντσέρτο. Παίρνει τα χρήματα για το κοντσέρτο μέσω εισιτηρίων. Πουλάει εισιτήρια. Μετά, γιατί αυτός ή εκείνη έχει το δικαίωμα πάρει και άλλα χρήματα μετά. Οδηγό του λεωφορείου. Και αυτό δεν παίρνει άλλα, άλλα χρήματα μετά γιατί οδηγούσε λεωφορείο. Είναι παράξενη συζήτηση, παράξενο θέμα. Ε, ζωγράφισα μια ζωγραφιά και αντεγράφει και παίρνω δικαιώματα. Γιατί? Το πούλησα. Πούλησα τον πίνακα. Πήρα τα λεφτά μου, τελείωσε. Έτσι δεν είναι. Πνευματικά δικαιώματα, ναι. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Αλλά είναι μεγάλο θέμα για συζήτηση. Δεν, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε στα πλαίσια που συζητήσαμε σήμερα με το deepfake κλπ. Στο Σαντιακό γίνεται ένα συνέδριο μεγάλο, η Comic στο Σαντιέγκο με εκατοντάδε καλλιτέχνε που πολλούν έργα τέχνη. Τα έργα του βασίζονται στα σχέδια κάποιου άλλου. Λέγεται fan Art. Μπορεί να αγοράσει τον Iron Man. Ε, με ακουαρέλα, με λάδι κλπ. Και, ρωτά τον καλλιτέχνη τι λέει η Marvel. Λέει η Marvel το δέχεται. Διότι είναι fan art. Βασίζουν οι καλλιτέχνες το έργο τους σε υφιστάμενο έργο κάποιο άλλο, ας πούμε στο, στην περίπτωση του Iron Man. Και λέγεται fan art. Σκεφτείτε το λοιπόν αυτό. Ίσως πηγαίνουμε πολύ μακριά με το copyright διαφορετικά. Υπήρχε άλλη ερώτηση που εκκρεμούσε. Μη φοβόσαστε λοιπόν με αυτά που έρχονται. Πρέπει να μάθουμε, να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, να έχουμε επίγνωση, να μην τα θεωρούμε σαν αληθινά, να πούμε εντάξει, Καλό αυτό, αλλά ξέρω εγώ, ίσως να είναι κάτι που δεν είναι αληθινό, ένα εφεύρημα. Μην δεχόσαστε ό,τι βλέπετε, με άλλα λόγια. Ασυζητητή και ανεξέλεγκτα. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω. Α, ορίστε, κύριε Μάτιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ε, προσκεκλημένους για τις ε, συναρπαστικές παρουσιάσεις τους. Ήταν συναρπαστικές και λίγο τρομακτικές θα έλεγα οι παρουσιάσεις. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει έναν διδάσκαλο. Ναι, ως διδάσκον μπορώ να πω ότι αν δώσω σε έναν υπολογιστή δεδομένα, ο υπολογιστής θα είναι πιο γρήγορος και θα γνωρίζει περισσότερα από μένα. Αυτό που δεν έχει όμως η τεχνητή νοημοσύνη είναι το πραγματικό συνέστημα, το οποίο είναι ανθρώπινο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Όταν βάλουμε σε έναν υπολογιστή ε, κάτι ε, το οποίο έχει φτερά, πούπουλα και, μια, και ένα ρίγχος, ε, ο υπολογιστής θα πει είναι πουλί. Μόνο ένα παιδί μπορεί να πει ότι είναι ο Ντάμπο το ελεφαντάκι. Υπάρχουν βέβαια περίπτωση μια μέρα οι υπολογιστέ να γίνουν απρόβλεπτοι και η κατάσταση τότε θα είναι τρομακτική. Ευχαριστώ. Ως μια τελική δήλωση. Ναι, θέλετε να πείτε κάτι κύριε Γκολτεβάη. Ναι, για το επίπεδο της γνώσης και της κατανόησης ήθελα να πω. Για παράδειγμα, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό. Η απόφαση δηλαδή που ένας άνθρωπος ε, θα πάρει και θα πει ε, θα πέσω πάνω στον άλλο άνθρωπο ή θα κάνω κάτι άλλο, θα γυρίσω αλλού το τιμόνι. Τι κάνω δηλαδή ως οδηγός, τι ξέρετε την κατάσταση αυτή. Η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται όλο και περισσότερο και κατανοεί τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα. Αυτό δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Και τα ρομπότ θα είναι όλο και πιο ανθρωποειδή. Μια μέρα πραγματικά θα είμαστε αντιμέτωποι με χαρακτήρες που δεν είναι πραγματικοί. Στη ζωή μας αυτό δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Απ' την άλλη όμως, υπάρχει και μια μεγάλη ευκαιρία μας από αυτό. Τώρα οι άνθρωποι είναι τυφλοί. Στο μέλλον θα βλέπουν, θα περπατούν χωρίς πόδια. Είναι πολλά τα τρελά που μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη για να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Όπως και το μαχαίρι μπορεί να κόψει ψωμί ή να δολοφονήσει. Είναι και τα δύο πάντοτε. Απλώς πρέπει κανείς να γνωρίζει και με την γνώση πάντα είναι ένα βήμα μπροστά. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι νομίζω. Ευχαριστώ. Να πω και μία λέξη στο τέλος. Πινόκιο ένα από τα παραδείγματα που πήραμε προηγουμένως. Αν δεν υπάρχουν σχόλια και κάποιος που να θέλει να μιλήσει, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτό το απόγευμα. Πήραμε εξαιρετικές πληροφορίες από όλους τους εμπειρογνώμονες. Μας δώσατε μια εικόνα για υλικό που μας ανανέωσε, μας εξέπληξε, μας τρόβαξε σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε αρκετό υλικό για να σκεφτούμε και να φτιάξουμε μια καλή έκθεση πρωτοβουλίας ως προς το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας δώσατε τα φώτα σας και φωτίσατε αυτό το σκοτάδι που κάποιοι από εμάς είχαμε σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω λίγο και στα γρήγορα ότι στις 16 Μαρτίου θα έχουμε την επόμενη συναδρίαση και παρακαλώ να προσέξετε ότι στις 2 Μαρτίου η συνεδρίαση έχει διαγραφεί. Ευχαριστούμε και τους ε, διερμηνείς. Όσοι δεν συμμετάσχουν, όσοι δεν θα συμμετάσχουν στη συνεδρίαση των συντονιστών, παρακαλώ να βγουν από την ένθουσα το συντομότερο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τους συντονιστές. Καλό απόγευμα.